Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Ας εγκρίνουμε γρήγορα την ημερήσια διάταξη. Εγκρίνετε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω ολόθερμα τον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ πέρα σήμερα για την τακτική αυτή ανταλλαγή απόψεων, τον οικονομικό διάλογο που προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία. Βέβαια, σήμερα η παρουσία σας εδώ μου δίνει τη δυνατότητα να σας ευχαριστήσω και να αποτίσω φόρο τιμής, θα έλεγα, σε εσά για τον πολύ σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραμετήσατε εδώ και πέντε χρόνια στη θέση του Προέδρου του Eurogroup. Ήσασταν πάρα πολύ κανός, ένας πολύ ισχυρός πρόεδρος του Eurogroup και συμβάλλατε στο να ληφθούν κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις και θα ήθελα να αποτίσω φόρο Τιμής στον τρόπο με τον οποίο συμβάλλατε στο να διαχειριστούμε τις πολύ δύσκολες συζητήσεις και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε για την Ελλάδα που συνέβαλαν τελικά στο να διατηρήσουμε την ενότητα της Ευρωζώνης. Θα έλεγα, λοιπόν ότι τα επιτεύγματα αυτά αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία της ε, δικής σας ε, πολύ σημαντικής ε, προσωπικότητας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για το έργο που επιτελέσατε και για την πολύ θετική συνεργασία που είχατε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, η σημερινή συνεδρίαση έχει μία πολύ συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, ένα πολύ συγκεκριμένο θεματολόγιο. Αλλά προφανώς να συγχαρώ και τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, τον Μάριο Σεντένο, ο οποίο εξελέγει πρόσφατα όπω το γνωρίζετε και ο οποίο θα αναλάβει το, αξίωμα του, το νέο του αξίωμα τον Ιανουάριο. Και προσβλέπουμε βέβαια σε μια θετική συνεργασία και με αυτόν και θα έχουμε επίση τη δυνατότητα ενδεχομένω να δούμε πώ θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία ανάμεσα στο Eurogroup και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην σημερινή συνεδρίαση επίση θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε την εφαρμογή των ειδικών αχώρα συστάσεων του 2017, καθώς επίσης και την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια ξέρετε ότι χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα, μια πολύ σημαντική δέσμη μέτρων, έκανε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση όσον αφορά το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Για μας λοιπόν θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό ακόμα περισσότερο, να υποβάλουμε σχόλια και παρατηρήσεις για αυτή τη δέσμη μέτρων και θα θέλαμε βέβαια να συζητήσουμε και για το ζήτημα αυτό με εσά, κύριε Γερούν Ντάισελμπλουμ. Θα έλεγα πάντω ότι οι χθεσινέ ανακοινώσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούν ένα σημαντικό ρώσιμο στην εμβάθυνση τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Κύριε Ντάισελμπλουμ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Με ιδιαίτερη χαρά επιστρέφω στην Επιτροπή Οικονομική και Νομισματική Πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την συνέχιση του οικονομικού μα διαλόγου αξιότιμα μέλη. Θα ξεκινήσω με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της χάραξης πολιτικής. Θα ήθελα καταρχάς όμως να αφαιρθώ στις οικονομικές μας προοπτικές. Ενώ συζητάμε σήμερα, η οικονομία της Ευρωζώνης είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό που ξεκίνησε ως εύθραστη ανάκαμψη του 2013 με πολλούς κινδύνους υποτίμησης, μετεξελίχθηκε σταδιακά σε στέρεα οικονομική ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής είχαμε 18 συναπτά τρίμηνα θετικής ανάπτυξης ε, του ΑΕΠΑ σε όλο ένα και πιο ευρία βάση και αυτό μας δίνει εμπιστοσύνη για το μέλλον. Εμπιστοσύνη η οποία αντικατοπτρίζεται και στη θετική στάση των καταναλωτών και των επενδυτών σε όλη την οικονομική περιφέρεια της Ευρωζώνης. Οι προβλέψεις του φθινοπόρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι οι οικονομικές προοπτικές θα παραμείνουν θετικές για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό αποτελεί βέβαια σημαντική μεταβολή σε σχέση με την αρχή αυτής της δεκαετίας, όταν εγώ έγινε επικεφαλής του Eurogroup δηλαδή, όταν το σύνολο της Ευρωζώνης και η ενότητα και κεραιότητα της Ευρωζώνης διέτρεχαν κινδύνους. Σίγουρα η Ευρωζώνη έχει ευνοηθεί από ούριους ανέμους, όπως το υψηλό επίπεδο νομισματικής διευκόλυνσης, αλλά νομίζω ότι αποτελεί αυτό και το αποτέλεσμα κάποιων πολύ δύσκολων μέτρων που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευρωζώνης και πιο συγκεκριμένα σε μεμονωμένα κράτη-μέλη. Καταφέραμε να διευθετήσουμε κάποια διαφορετικά ζητήματα και βέβαια αυτό οδήγησε σε κοινωνικό αλλά και πολιτικό κόστος. Αλλά όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σημαντικά θετικά αποτελέσματα στις χώρες μου. Ως προς αυτό θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στην Ελλάδα. Από την αρχή του τρίτου προγράμματος της, στα πλαίσια του ESM, το καλοκαίρι του 2015, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει ένα εντυπωσιακό και ευρύ κατάλογο σημαντικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, όσον αφορά τον εξυγχρονισμό της αγοράς εργασίας και προϊόντων. Βέβαια, ακόμα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, αλλά πάντως σίγουρα η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα από πολιτικής και οικονομικής πλευράς. Και αυτό μας έχει επιτρέψει να ολοκληρώσουμε επιτυχώς την τρίτη αξιολόγηση. Όπως ξέρετε, οι αρχές και τα θεσμικά όργανα κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο όσον αφορά τους επικυροποιημένους όρους οικονομικής πολιτικής. Επομένως, η Ελλάδα τώρα θα πρέπει να εφαρμόσει μια σειρά προαπαιτούμενων δράσεων οι περισσότερες εκ των οποίων θα εφαρμοστούν πριν τα Χριστούγεννα και οι υπόλοιπε στις αρχές Ιανουαρίου, έτσι τουλάχιστον έχω ενημερωθεί. Και εφόσον όλα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, το Eurogroup θα είναι λογικά σε θέση στην επόμενη συνεδριασή του 22 Ιανουαρίου να εγκρίνει μία ακόμα εκταμίευση δόσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Το Eurogroup επίσης αποφάσισε τον Ιούνιο να ξεκινήσει από το 2018 την τεχνική εργασία για το ζήτημα των μέτρων για το χρέος. Όπως ξέρετε, ο ESM αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει να εφαρμόσει μια σειρά από βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τα οποία θα βοηθούσαν βέβαια την Ελλάδα, αλλά ήδη από τον ε, Ιανουάριο θα είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε περισσότερα μέτρα για να βοηθήσουμε την ανάκαμψη της Ελλάδας και για να καταφέρουμε και μεσοπρόθεσμα να στηρίξουμε την εξυπηρέτηση του χρέους στην Ελλάδα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ καλά νέα, πολύ θετικές εξελίξεις και ουσιαστικά θα βοηθήσουν την Ελλάδα να βγει από το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018. Τα όσα ισχύουν για την Ελλάδα ισχύουν κατά κάποιο τρόπο και για το υπόλοιπο της Ευρωζώνης. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε δύσκολες επιτυχίες, αλλά πολλά πράγματα ακόμα απομένουν να γίνουν στο μέλλον. Ξέρετε ότι είμαι αισιόδοξο. Κάποιος εδώ πέρα με έχει αποκαλέσει στα πλαίσια της Επιτροπής σας τον πιο αισιόδοξο στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Ξέρω όμω ότι έχουμε πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα στην Ευρωζώνη και ότι έχουμε ακόμα σημαντικά πράγματα να κάνουμε στο μέλλον. Τώρα, η δημοσιονομική πολιτική στα πλαίσια τη Ευρωζώνης συζητήθηκε και αυτή τη Δευτέρα στα πλαίσια των δημοσιονομικών προγραμμάτων των σχεδίων προπολογισμού των χωρών της Ευρωζώνης. Εμείς στο Eurogroup συμφωνήσαμε ουσιαστικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται ένας εν γέννη ουδέτερος δημοσιονομικός προσανατολισμός για το σύνολο της Ευρωζώνης στα πλαίσια της τρέχουσας συγκυρίας. Αλλά βέβαια εφίστανται ακόμα διαφορές μεταξύ των κρατών και δεν μπορούμε να πούμε ότι η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια ενιαία προσέγγιση για όλες τις χώρες. Μόνο λίγες χώρες διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν για επιπλέον επενδύσεις ή δαπάνες που θα ευνοούσαν την παραγωγικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε στα σχέδια προπολογισμού έξι χωρών ότι διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωση με του δημοσιονομικού κανόνε. Και αυτό περιλαμβάνει χώρε που έχουν ε, ακόμα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέου. Οι χώρε αυτέ θα πρέπει να κάνουν κάθε το δυνατό προκειμένου να συμμορφωθούν με το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσουν μια ακριβοδίκαιη εφαρμογή των κανόνων. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το προληπτικό σκέλος του συμφώνου και να χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο του χρέους στα πλαίσια της δημοσιονομικής εποπτείας. Πέρα όμω από τι υγιεί δημοσιονομικές πολιτικέ, οι χώρε θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει, προκειμένου επιχειρηματίες, επενδυτές, νέοι και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι να έχουν ε, σημαντικές ευκαιρίες ε, να συμμετάσχουν στην οικονομία και να ενισχύσουν έτσι την οικονομία. Γι' αυτό το λόγο στα πλαίσια του Eurogroup αφιερώσαμε αρκετό χρόνο διεξάγοντα τις λεγόμενες θεματικές συζητήσει για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δηλαδή τη δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα για τα ζητήματα αυτά. Ασχοληθήκαμε με τη φορολογική επιβάρυνση τη εργασία. Το ζήτημα αυτό μας απασχόλησε και την προηγούμενη Δευτέρα και πολλά κράτη-μέλη έχουν αναλάβει μέτρα προκειμένου να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, ιδίως για το χαμηλότερο λεγόμενο τμήμα τη αγορά εργασία. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την έμπρεθμη λειτουργία των αγορών εργασία και μπορεί να δώσει νέε ευκαιρίε στου πολίτε προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία, να βρουν μια θέση απασχόληση και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν οι πολίτε να έχουν και υψηλότερε αποδοχέ στα πλαίσια τη αγορά εργασία. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα αυτό επί το οποίο θα πρέπει από κοινού όλοι να συνεργαστούμε, μολονότι βέβαια το ζήτημα αποτελεί σαφώ εθνική αρμοδιότητα, θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό μπορούμε και θα πρέπει από κοινού να το προωθήσουμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια άσκησα πίεση και αυτό ελπίζω ότι θα γίνει και στο μέλλον να έχουμε κοινά πρότυπα, ποιοτικά, κοινού δείκτε συγκριτική αξιολόγηση, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα κοινό υψηλό επίπεδο στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Α περάσουμε τώρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την Τραπεζική Ένωση. Η Ευρωζώνη προφανώς χρειάζεται έναν εύρυθμο τραπεζικό τομέα. Οι τράπεζες θα πρέπει να εξυπηρετούν τις επιχειρήσει και θα πρέπει βέβαια να ισχύουν ισότιμοι κανόνε για όλε τι τράπεζε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την εργασία για μια ολοκλήρωση τη τραπεζική Ένωση. Η εργασία αυτή προφανώ έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται ακόμα και αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε κάποια ενθαρρυντικά παραδείγματα τη εργασία που γίνεται στην Ισπανία και στην Ιταλία και θα μπορούσαμε να λύσουμε διδάγματα από τις πρόσφατες ε, περιπτώσεις ε, εξυγίανσης ε, των τραπεζών ή αναδιάρθρωση των τραπεζών και αυτό συμβάλλει με τη σειρά του στην ολοκλήρωση Τραπεζικής Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στην ευάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το Eurogroup προετοίμασε τη σύνοδο κορυφή τη Ευρωζώνη που θα λάβει χώρα στι 15 Δεκεμβρίου. Αυτό έγινε σε σύνθεση ανοιχτή και στα 27 κράτη-μέλη, ακολουθώντα την αρχική πρωτοβουλία του Προέδρου Τούσκα ασχοληθήκαμε με τρία βασικά ζητήματα στις τρεις βασικές συζητήσει προπαρασκευαστικές που είχαμε του τελευταίου μήνες. Ασχοληθήκαμε καταρχάς με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, εν συνεχεία με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωση και τέλος με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Οικονομική και Νομισματικής Ένωση στο πλαίσιο του οποίου θα μπορούσαμε να δούμε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αν επαρκεί, αν είναι κατάλληλο, αν θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Και είπαμε ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένω να χρησιμοποιήσουμε και νέα εργαλεία, νέα μέσα δημοσιονομική πολιτική. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο συζητήσαμε τα θέματα αυτά μεμονωμένα και ξεχωριστά, ενώ τη Δευτέρα κάναμε μια οριζόντια συζήτηση προκειμένου να ακούσουμε ποιε είναι οι προτεραιότητε των συναδέλφων από τι διάφορε χώρε και πώ θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Εγώ σε σχέση με αυτό θα κάνω μια παρουσίαση στη Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωζώνη. Θα ήθελα απλώ να σα πω Ποιε εντυπώσει έχω αποκομίσει μέχρι στιγμή όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, υπάρχει μια ευρεία συνένεση ότι η Ευρωζώνη θα πρέπει να βασιστεί στην ε, εμπειρία που έχει στη διαχείριση των προγραμμάτων προσαρμογή και να βαθμίσει περισσότερο το ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα. Κατά συνέπεια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα έχει ένα μικρότερο ρόλο στο μέλλον και υπάρχει ευρεία υποστήριξη στην Ευρωζώνη για να διατηρήσουμε την υφιστάμενη θεσμική δομή του ESM. Υπάρχει πλέον μια ευρή εμπιστοσύνη των κρατών μελών προς τον μηχανισμό αυτόν. Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα ρόλο για να σημειώσουμε πρόοδο στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Βασιζόμαστε στον συμφωνημένο δικό χάρτη, συμφωνήθηκε το 2016 στα πλαίσια του Συμβουλίου όπου προβλέπεται μείωση του κινδύνου αλλά και επιμερισμός του κινδύνου με μια ισορροπημένη προσέγγιση και ω προ τα δύο. Θα πρέπει και στου δύο αυτού τομεί, μείωση του κινδύνου και επιμερισμό του κινδύνου, να σημειώσουμε ισορροπημένη πρόοδο και θα μπορούσαμε εδώ πέρα να προωθήσουμε περισσότερο την δέσμη μέτρων την οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία θα πρέπει να σαν αντικείμενο περαιτέρων διαπραγματεύσεων. Και θα πρέπει βέβαια να ασχοληθούμε και με κάποια ζητήματα όπω τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για τα οποία θα πρέπει να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να λάβουμε πιο σημαντικά βήματα, πιο σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά το ζήτημα του επιμερισμού κινδύνου σε ζητήματα όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας των Καταθέσεων ή το κοινό προστατευτικό σύστημα για το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Στόχος του Προέδρου Τούσκ είναι να φτάσουμε σε πιο σημαντικές αποφάσεις σε μια άλλη σύνοδο της Ευρωζώνης που θα λάβει χώρα τον ε, Ιούνιο του 2018 και θεωρώ ότι θα είναι δυνατό στα πλαίσια της μελλοντική αυτή συνόδου να σημειώσουμε πρόοδο για τα ζητήματα αυτά. Όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο τη ΟΝΕ, υπάρχει μια γενικότερη συνένεση ότι όντω ε, το πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, μερικές φορές προβληματικό. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να διατηρήσουν την εθνική κυριότητα για την ΟΝΕ και θα πρέπει προφανώς ο τρόπος λειτουργίας της ΟΝΕ να απλουστευθεί. Τώρα, οι συζητήσεις για κάποια νέα δημοσιονομικά μέσα και εργαλεία έχουν προχωρήσει λιγότερο. Ακούσατε και από τον Πρόεδρο ότι είχαμε χθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία ανακοίνωση για νέα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα όμω δεν έχει καταλήξει σε μία συγκεκριμένη απόφαση. Αναφέρθηκε ενδεχομένω σε έξι διαφορετικά μέσα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Και βέβαια, αν πρέπει όλα αυτά να ενταχθούν στο γενοτικό προπολογισμό, τότε η επόμενη συζήτηση που θα γίνει για το στο νομικό πλαίσιο θα είναι για να το θέσω οικός ιδιαίτερα δύσκολη. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια θα είναι τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον, πώς θα σχεδιαστούν αυτά, πώς θα χειριστούμε, πώς θα χρηματοδοτηθούν, από πού θα έρθουν τα χρήματα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στο μέλλον να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα ζητήματα προκειμένου να προετοιμάσουμε τις νέες αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε τον Ιούνιο. Βέβαια έχουμε ένα πολύ θετικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ήδη τη Δευτέρα οι επαφές που κάναμε ήταν πολύ θετικές. Δεν είχαν γίνει τότε ακόμα οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι οι προτάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα περιεκτικές. Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις όσον αφορά τα δημοσιονομικά ζητήματα, αλλά και όσον αφορά το ζήτημα της ε, διακυβέρνησης. Ορισμένα ζητήματα θα πρέπει άμεσα να τα προωθήσουμε, αλλά πάλι θα πρέπει να τα συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Εν κατακλείδη, θα έλεγα ότι ε, η υφιστάμενη οικονομική συγκυρία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για μας. Έχουμε πλέον μια νέα δυναμική στη συζήτηση που γίνεται για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ο πρόεδρος Μακρόν έχει συμβάλει σε αυτό. Το Brexit το δικό του τρόπο επίσης, καθώς επίσης και η στάση της Αμερικανικής κυβέρνησης, ενδεχομένως χωρίς να το θέλει, αφελά της. Νομίζω πάντως ότι ε, τώρα και τους επόμενους έξι μήνες θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο στη συζήτηση αυτή για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις τον Ιούνιο. Εγώ δεν θα συμμετέχω βέβαια πλέον σε αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κοιτώντας λίγο τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι ζήσαμε αρκετά δύσκολες στιγμές στα πλαίσια της Ευρωζώνης, στα πλαίσια της οικονομίας μονομένων κρατών μελών και βλέπουμε ακόμα τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης. Προφανώ λοιπόν τα πράγματα δεν είναι ακόμα τέλεια, πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν ακόμα. Εγώ προσπάθησα να συμβάλλω προκειμένου να διατηρήσω την ακαιρεότητα και την ενότητα τη Ευρωζώνη και προκειμένου να βγούμε από την κρίση πολύ πιο ισχυρή και δυνατή. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει και αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική στέρεη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να βασιστούμε και τι πολιτικέ μα εργασίε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοδηματική αυτή συνεργασία που είχαμε και εγώ άγγλισα πάρα πολλά διδάγματα και έμαθα από τι επαφέ που είχα μαζί σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τη συνεργασία συνεργασία που Ευχαριστώ πολύ, Γερούν, και αυτό δείχνει νομίζω πως ολόκληρη η Επιτροπή ε, σε συγχαίρει για την πολύ σημαντική συμβολή σου για το μέλλον και για το μέλλον βεβαίως σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία και τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Κύριε Βάλτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντάισελμπλουμ. Τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος του Eurogroup ε, ζήσατε κι εσείς ε, κάποιες ε, έντονες και τραχώδεις στιγμές για την Ευρωζώνη, τις οποίες επίσης ε, συνδιαμορφώσατε. Θα ήθελα λοιπόν και εξ ονόματος του ΕΛΚ να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας. Συνεισφέρατε στην σταθερότητα των χωρών της Ευρωζώνης και θα έλεγα μάλιστα ότι καταφέρατε να ωφελήσετε την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση οικονομικής ανάπτυξης. Ε, έχουμε λοιπόν ανάπτυξη και οι προγνώσεις της Κομισιόν για το επόμενο έτος είναι θετικές, ε, κατά το οποίο οφείλεται και στις ε, διαρθρωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών όμως Οπωσδήποτε η δουλειά μας τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι απλή. Οι τελευταίες προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ε, και για θεσμικές εξελίξεις ε, αφορούν ιδιαίτερα την Ευρωζώνη. Αναφέρατε ότι την Δευτέρα συζητήσατε αυτές τις προτάσεις με την Κομισιόν στο Eurogroup και εμείς βεβαίως ε, θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό και θα θέλαμε να ρωτήσουμε την Κομισιόν γιατί έγινε στο Συμβούλιο και όχι στο Κοινοβούλιο αυτό. Οπωσδήποτε ως ομάδα του ΕΛΚ η πρόταση αυτή να αλλάξει ο μηχανισμός σταθερότητας σε ένα ευρωπαϊκό δουνουτού είναι κάτι το οποίο α, ακούσαμε. Θα πρέπει όμως να υπάρξει μία συζήτηση εκτεταμένη επί του θέματος και να δούμε βεβαίως και τις πιθανές αρμοδιότητες του προτινόμενου Υπουργού Οικονομικών της Ευρωζώνης που θα προεδρεύει και στο Eurogroup. Αυτά βεβαίω ε, τα βλέπουμε σε σχέση με κάποιες δύο οργανικές δικλείδες ασφαλείας. Η ερώτησή μου λοιπόν για εσάς σήμερα είναι πώς αξιολογείτε τις προτάσεις της Κομισιόν για τις αρμοδιότητες του δικού σας ε, αξιώματος ε, το οποίο εγκαταλείπετε τώρα και που βλέπετε τις δυνατότητες συγκρούσεων ε, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Πρόεδρου του Ευρωγκρουπ και του Επιτρόπου Αρμοδίου για τα Οικονομικά. Σας ευχαριστώ κύριε Μπάλτς για τα καλά σας λόγια. Να συνεχίσω στα, αγγλικά για να μην μπλέξω τώρα με τα γερμανικά. Η Κομισιόν δεν παρουσίασε τις προτάσεις της στο Eurogroup έτσι για να σας διορθώσω ως προς αυτό. Ε, γνωρίζαμε χοντρικά τις προτάσεις βεβαίως γιατί είχαμε τις ομιλίες του Προέδρου Γιούνκερ στο Κοινοβούλιο οπότε εσείς ενημερωθήκατε πρώτοι. Ε, είπα μία φορά να υπερασπιστώ και την Κομισιόν. Η ΔΕ Κομισιόν τώρα στι προτάσει τη μιλάει για Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών, όχι μόνο για την Ευρωζώνη. Οπότε έχει πολύ εκτεταμένε και ευρύτατε ιδέε. Αλλά επίση πολύ ασαφής σε κάποια στοιχεία. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τις δημοσιονομικές πολιτικές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωζώνη. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Όπως ξέρετε το σύνολο των εθνικών προϋπολογισμών είναι 50 φορές το μέγεθος του προϋπολογισμού της Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι ένας Υπουργό Οικονομικών της Ένωσης θα ελέγχει τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Θα είναι ένα τεράστιο βήμα, αλλά γύρονται και τεράστια ζητήματα πολιτικής, συνταγματικά ζητήματα, δημοκρατικής νομιμοποίησης, αν έχει κάποιος τέτοια άμεσο έλεγχο του προπολογισμού, πρέπει να ελέγχει και που δαπανώνται. Αλλά ε, γύρω στο 80% του προπολογισμού στη χώρα μου πηγαίνει σε κοινωνική ασφάλιση, συντάξεις, ε, υγεία και εκπαίδευση. Αυτά όμως είναι αρμοδιότητες των εθνικών κυβερνήσεων, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ο έλεγχος του προϋπολογισμού θα πάει σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να δούμε αυτούς τους τομείς πολιτικής. Είναι λοιπόν μεγάλη συζήτηση. Και πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς όταν μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις και είναι θετικό το ότι η Κομισιόν έχει κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο για τον ρόλο ενός Ευρωπαϊκού Οικονομικών, αλλά γύρει πολλά ερωτήματα τα οποία αφήνει αναπάντητα. Ρεαλιστικά μιλώντας λοιπόν, το Eurogroup θα επιμείνει στο να έχει δικό του πρόεδρο. Μόλις ε, κλέξαμε τον Μάριο Σεντένο για δυόμιση χρόνια και υπάρχει αίσθηση στο Eurogroup ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ του ρόλου του Eurogroup που είναι διακυβερνητικό και της Κομισιόν η οποία είναι θεματοφύλακας των συνθήκων για α, όλους μας, για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μείνω σε αυτά γιατί μπορούσα να πω πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ. περβάνω Περές. Ευχαριστώ. Στο όνομα τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε. Θυμούμε πάρα πολύ καλά πότε αναλάβατε, όταν γινόταν ε, χαμός στην Ελλάδα και αναλάβατε την έξοδο από την κρίση, τη διαχείριση της κρίσης και μάθαμε μαζί σας ε, τα αποτελέσματα. Είσαστε ένας ε, αναμφίβολα από που καλύτερα διαχειρίστηκαν και γνώρισαν την ε, κρίση μπόρεσατε να διαχειριστείτε τις σχέσεις και με το Δουνουτού και σας εύχομαι, ε, εύχομαι μάλλον διευρυμένη επιτυχία με βάση τις δικές σας επιτυχίες στον διάδοχό σας. Μιλήσατε για την ε, ουδέτερη ομαδοποιημένη νομικό ε, προσανατολισμό. Ε, λοιπόν, νομίζω πως είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο και χρησιμοποιείται στο ΕΚΟΦΗΝ. Το θέμα δεν είναι να, να παρατηρούμε ποια είναι η ομαδοποιημένη κατάσταση, αλλά να χρησιμοποιήσουμε αυτό το, τα στοιχεία ως εργαλείο για να ασκήσουμε μια αντικυκλική πολιτική εκεί όπου πρέπει. Διερωτώ με σε ποιο βαθμό εσείς συμμερίζεστε αυτή την προσέγγιση. Έπειτα, Αναφερθήκατε στα ερωτηματικά που υπάρχουν μέσα και στο Eurogroup σε σχέση με τη λειτουργία ενός προπολογισμού της Ευρωζώνης. Όμως πιστεύω υπάρχει ένα στοιχείο, μια ιδέα επί της οποίας υπάρχει συνένεση, ότι δηλαδή χρειάζεται στην Ευρωζώνη μια λειτουργία σταθεροποίησης. Όμως πρέπει να εκφράσω την ε, απογοήτευσή μου για τη δέσμη μέτρων ε, που ε, υιοθετήθηκε χθε και συμμερίζομαι και τις επικρίσεις του συναδέλφου Μπάλτ. Δεν καταλαβαίνω πώς η Κομισιόν δεν βρήκε τον τρόπο να υποβάλει εδώ ενώπιον του Κοινοβουλίου πριν ή μετά αυτές τις προτάσεις. Είναι μια άρνηση διαλόγου με τους εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών που είναι δικαιολόγητη. Για ε, αυτή τη σταθεροποίηση το κληροδότημα που αφήνεται στον διάδοχό σας ε, ε, δεν είναι κατά τη γνώμη σας επίγον το να δημιουργηθεί ένα τέτοιο εργαλείο ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η λειτουργία. Τρίτη ερώτηση, σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση για την οποία κάνατε πολύ λόγο. Και αναφέρετε αυτή την ιδέα της εξισορρόπησης ανάμεσα στο risk sharing και στο risk reduction. Αμοιβοποίηση δηλαδή του κινδύνου και μείωση του κινδύνου εμείς προσπαθούμε με την εποπτεία και τα λοιπά, θύνοντες προσπαθούν να οργανώσουν την ε, τραπεζική αναδιάρθρωση όσον αφορά το risk reduction. Αλλά μήπως θα έπρεπε να προχωρήσουμε και στο περισσότερο λίγο στο risk reduction συνεχίζοντας την εργασία ε, και για το άλλο πακέτο. Αν όμως δούμε τη ζυγαριά, έχουμε μια αντίληψη μιας νέας, ενός νέου είδους ε, φυσικής Δηλαδή, ότι πρώτα θα πρέπει να έχουμε κατεβάσει κάτω-κάτω το ένα κομμάτι της ζυγαριάς πριν αρχίσουμε λίγο να βαραίνουμε και στο άλλο. Και βέβαια αν έχετε κάποια ιδέα για το τι θα κάνετε από εδώ και μπρος στα διαδρομία σας, πολύ θα θέλαμε να το γνωρίζουμε. Ευχαριστώ κυρία Μπερές. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια. για την ε, κοινή αυτή για το κοινό αυτό δημοσιονομικό εργαλείο για την Ευρωζώνη το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια αντικυλική πολιτική αυτό είναι γεγονός αλλά το πώς θα γίνει στην πράξη είναι ένα θέμα γιατί ακόμα Ε, οπωσδήποτε στα χρόνια της ε, κρίση, τώρα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα είχαμε τεράστιε διαφορέ μεταξύ των χωρών που είχαν ανάπτυξη μια πολύ μεγάλη χώρα είχε και ικανό πλεόνασμα και μπορούσαμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη χώρα να ασκήσει αντικυκλικές πολιτικές ε, για να γίνει αυτό θα έπρεπε να κάνει λιγότερες δαπάνες. Σε άλλες χώρες δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο και η οικονομία ακόμα είναι πολύ ασθενείς και οι χώρες αυτές ε, θα χρειάζονταν περισσότερες δημοσίες επενδύσεις. Δεν έχουμε λοιπόν τα μέσα για να το αντισταθμίσουμε αυτό. Και έτσι ερχόμαστε ε, στο άλλο θέμα του να έχουμε μια δημοσιονομική ικανότητα ή ένα εργαλείο σταθεροποίησης για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Η Κομισιόν έχει φορές, ε, πολλές και διάφορες ιδέες στις προτάσεις της το κάνουν αυτό μάλλον γιατί γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει συμφωνία και σύγκληση ιδεών οπότε αφήνουν στο πακέτο όλες τις διαφορετικές ιδέες μιλάνε για ένα εργαλείο το οποίο θα ενισχύσει και θα στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να υπάρχουν και αν θα πρέπει να είναι μεταφορές ή ε, χρηματοδότηση η οποία θα εξοφληθεί μετά. Και βεβαίως το εάν θα προέρχεται από τον κοινοτικό υπερπολογισμό ή από κάποιο άλλο μέσο, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή κάποιο άλλο φορέα της Ευρωζώνης. Βεβαίως υπάρχει και το μέσο σύγκλησης. Ε, μπορεί βεβαίως να πει κάποιος πως τα διαρθρωτικά ταμεία ήδη παρέχουν αυτή τη στήριξη για τη σύγκληση και μετά έχουν και άλλες ιδέες για το μέσο σταθεροποίησης, ε, επιδόματα ανεργίας, ε, αντασφάλιση και ένα σύστημα προστασίας επενδύσεων. Όλα αυτά δείχνουν ότι είμαστε ακόμα στην αρχή της ε, συζήτησης. Προσωπικά θεωρώ ότι ένα μέσο σταθεροποίησης χρειάζεται για δυσμενή σοκ και αναταράξεις σε συγκεκριμένα κρατημέλη για να στηριχθούν αυτά ειδικά για τις ε, χώρες της Ευρωζώνης θα έπρεπε να γίνει με τη μορφή ενός χρηματοδοτικού μέσου αντί για α, μεταφορές ε, κονδυλίων και βεβαίως θα έπρεπε να υπάρξουν και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να δούμε και να αντιμετωπίσουμε και τις αιτίες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη τώρα το τι θα γίνει. Τέλος, μιλήσατε για την μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ναι, το τελευταίο έτος, εξάμεινο, δουλεύουμε μόνο, υπήρξε δουλειά μόνο στη μείωση του κινδύνου και όχι στον διαμοιρασμό του. Βεβαίως ε, ξεκίνησε κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. ξεκίνησα με το Ταμείο Διάσωσης, το οποίο θα έλεγα ότι μοιράζει τον κίνδυνο, οπότε είναι κάπως μοιρασμένα τα πράγματα. Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτό που λένε κάποιοι συναδελφοί μου ότι θέμε περισσότερο από αυτό πριν κάνουμε το άλλο. Αυτό είναι δικαιολογία για να μην κάνουμε τίποτα τελικά. Και ε, το, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να προχωρήσουμε και στα δύο όχι να λέμε όλο το ιστορικό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να τα να αντιμετωπίσουμε πριν μιλήσουμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης ε, καταθέσεων. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι σε κάποιες ε, χώρες ένα τέτοιο σύστημα εγγύησης καταθέσεων είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Μάλιστα. Οπότε θα έλεγα ότι πρέπει να συνεχίσουμε την πρόοδο και στα δύο μέτωπα και να μην μπούμε σε παιχνίδια λέξεων. Τέλος, ρωτήστε για το δικό μου το μέλλον. Είπα αστειευόμενος στον πρόεδρο ότι ίσως θα πρέπει να είμαι ο πρώτος που θα εκμεταλλευτώ το ευρωπαϊκό επίδομα ανεργίας, αλλά ελπίζω όχι, για προσωπικούς λόγους. Τίποτα συγκεκριμένο λοιπόν δεν έχω να σας πω ως προς αυτό. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς. Ε, κύριε Ντάισεμπλουμ, κύριε Ντάισεμπλουμ, ε, αναφερθήκατε, αναφερθήκατε στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι έχετε επιλεκτική μνήμη. Ξεχάσατε να μας πείτε ότι η φτώχεια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι στο 40%, ότι το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25%, ότι η ανεργία είναι τώρα κοντά στο 20% αλλά έχει φτάσει στο 26%, ότι οι συντάξεις μειώθηκαν 40%, ότι μειώθηκαν οι μισθοί. Επομένως, θα περίμενα στην τελευταία σας συνεδρίαση εδώ, στην παρουσία σας, θα είχατε μια ευκαιρία να κάνετε και μια αυτοκριτική, διότι το πρόγραμμα, τα μνημόνια απέτυχαν στην Ελλάδα. Ο ίδιος ομολογήσατε πρόσφατα ότι διασώθηκαν οι τράπεζες και όχι η ελληνική οικονομία και θα περίμενα να ζητήσετε και ένα μεγάλο συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και κυρίως από τα εκατομμύρια των ανέργων. Η ερώτηση όμως που θα σας θέσω αφορά τα κόκκινα δάνεια. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με το τρίτο πρόγραμμα έχει, πάρει, έχει συμφωνηθεί να πάρει 86 δισεκατομμύρια ευρώ δάνειο. Όμως, σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Ρέγκλιν, θα περισσέψουν 25 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του προγράμματος. Επομένως η πρόταση που θέτουμε είναι η εξής. Ένα ποσό από αυτά, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός ταμείου σωτηρίας για κόκκινα δάνεια. Ένα ταμείο διαχείρισης των κόκκινων δανείων, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί φτωχοποιημένοι Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους, δεν είναι κακοπληρωτές, απλά επειδή είναι άνεργοι, επειδή έχουν χαμηλά εισοδήματα πλέον, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτό το Ταμείο για Κόκκινα Δάνεια θα μπορούσε στην ουσία να στηρίξει την αγορά δανείων περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ στεγαστικά δάνεια, διότι στο 10% προτίθενται να ταρπάξουν τα distress funds. Επομένως η ερώτησή μου είναι πρώτον, συμφωνεί το Eurogroup να διατεθεί ένα ποσό για τη δημιουργία ενός ταμείου σωτηρίας για κόκκινα δάνεια και δεύτερον να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο οι δανειολήπτες θα μπορούν να κατά προτίμηση να αγοράσουν το δάνειό τους στην τιμή πρώτης προσφοράς που κάνουν τα distress funds. Αυτή την ίδια ερώτηση την έθεσα και στον κύριο Ντράγκη εδώ πριν 15 ημέρες και με παρέπεμψε στο Eurogroup. Το Eurogroup υποτίθεται ότι είναι αυτό που δανειοδοτεί την Ελλάδα. Επομένως συμφωνείτε ένα μέρος των χρημάτων που υπολείπονται από το δάνειο να δοθούν για τη δημιουργία ενός Ταμείου Σωτηρίας για κόκκινα δάνεια. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, Ειλικρινά, Πρόεδρε, μόλις ξεκίνησε η ομάδα εργασίας για την Τραπεζική Ένωση, με τον ε, κεντρικό διαπραγματευτή της Κομισιόν και τα στοιχεία είναι αρκετά ενθαρρυντικά για το πώς προχωράει η, Ευρωπα... η ελληνική οικονομία στους διάφορους τομείς. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, τα στοιχεία είναι όντως πολύ ενθαρρυντικά και για την μείωση των ε, δανείων και αυτή η διαδικασία ξεκινά. Λέτε πως έχω επιλεκτική μνήμη. Αντίθετα έχω πολύ καλή μνήμη. Και δεν δέχομαι αυτή τη γραμμή σκέψης που ακούω συχνά ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα προκάλεσαν τα προβλήματα στην Ελλάδα. Δεν το δέχομαι απλούστατα. Και μάλιστα η μνήμη μου θυμάται και πριν ε, ξεκινήσει η κρίση εκείνα τα χρόνια και πόσο ευάλωτες οι χώρες μας ήταν και πόσο ευάλωτες μπήκαν στην κρίση ε, και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Οι κίνδυνοι ε, χτίζονταν μη παραγωγικές επενδύσεις, τεράστια λάθη που διαπράχθησαν τα χρόνια πριν την κρίση. Αλλά έχετε δίκιο ότι έγιναν και λάθη μετά την έναρξη της κρίσης, στο πώς αντιδράσαμε και νομίζω πρέπει να είμαστε ειλικρινεί όταν λέμε ότι τα πρώτα χρόνια και σίγουρα στο πρώτο, στα πρώτα προγράμματα ε, αυτοσχεδιάσαμε σε μεγάλο βαθμό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίσαμε τις τράπεζες ήταν πολύ δαπανηρός και όχι αποτελεσματικός αρκετά. Ο κόσμος μας επικρίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσαμε τις τράπεζες στην Ελλάδα στην πρώτη φάση στην ουσία έσωσε τους επενδυτές που ήταν εκτός Ελλάδας βασικά. Αυτό είναι αλήθεια νομίζω και γι' αυτό και είμαι υπέρ των νέων κανόνων BRD και την αρχής του «Μπέιλιν» γιατί δεν νομίζω ότι θα πρέπει ξανά να διασώσουν επενδυτές που θα έπρεπε να έχουν φροντίσει καλύτερα να καλύψουν τους, δικούς, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Αυτό ήταν ένα λάθος λοιπόν που έγινε στην αρχή της κρίσης. Είναι εύκολο να λέει κανείς και ίσως είναι ε, παλιά μου γνώση να σε είχα πρώτα. Αλλά και εγώ αν ήμουν εκεί από την αρχή θα έπρεπε να αυτοσχεδιάσω. Ήταν μια τεράστια κρίση, τεράστια κίνδυνη διάδοση και πλήρους κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λοιπόν, ήταν τέτοιε οι περιστάσει όταν λήφθησαν αυτέ οι αποφάσει και άφησαν πολλέ από τι χώρε μα με πολύ ψηλό χρέο και γρήγορα και απαιτητικά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Αυτή είναι η αυτοκριτική μου. Ελπίζω τώρα να τα καταφέρνουμε πολύ καλύτερα και, ε, και στο τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα συμβαίνει κάπου το ίδιο. Από τα 86 δις είχαμε 25 για την αναποκεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αλλά λόγω του πώς γίνεται τώρα δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Έχουμε χρησιμοποιήσει 4,5 δις μόνο, γιατί μεγάλο κομμάτι της λύσης ευρέθη από ιδιώτες επενδυτές και πρέπει να βάλουμε μόνο ένα πολύ μικρότερο ποσό δημοσίου χρήματος στις τράπεζες. Και από εκεί προκύπτει η ερώτησή σας, τι θα κάνουμε με τα χρήματα που περίσεψαν. Μα δεν περίσεψαν, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, μπορείτε να τα δαπανίσετε για κοινωνικούς σκοπούς για και δημόσιες επενδύσεις και όλα αυτά θα μπορούσατε να τα χρησιμοποιήσετε, αλλά δεν έχουν περισσέψει, προστίθενται στο χρέος της Ελλάδας. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αποπληρωθούν. Θα βαρύνουν ακόμα περισσότερο το χρέο. Δεν είναι τζάμπα λεφτά. Ας είμαστε ακριβείς. Ε, τα κόκκινα δάνεια τώρα. Ε, έχουμε μιλήσει για μια εξέβρεση μιας λύσης ε, ιδιωτικής και ε, όντω δεν θα πρέπει οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τι τράπεζε και του επενδυτέ. Από την άλλη πλευρά, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολύ ευάλωτου ανθρώπους ε, που πήραν δάνεια κτλ. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορείς να κάνεις και που γίνονται και στην Ελλάδα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι εκείνη τα θύματα των πληστηριασμών των ε, κόκκινων δανείων που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέσο ώστε οι τράπεζε να σταθούν πάλι στα πόδια τους, να καθαρίσουν τους ολολογισμούς τους και θα έπρεπε παράλληλα να υπάρχουν πολιτικές ώστε να προστατευτούν οι ευάλωτοι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαι βέβαιος ότι πρέπει να υπάρχει τέτοιο τεράστιο ταμείο γιατί και αυτό πάλι από του φορολογούμενου θα πληρωθεί. Wolfgang Klintz. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Μου κάνει εντύπωση το ότι ο τραπεζικός τομέας παραμένει κατακαιρματισμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη πιο συγκεκριμένα. Μολονότι έχουμε πλέον ένα ενιαίο νόμισμα και μολονότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για την ένωση των κέφαλα αγορών. Κατά την άποψή σας λοιπόν, για ποιο λόγο ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν είναι πλέον πιο ενοποιημένος πανευρωπαϊκά. Πιστεύετε εσείς ότι θα αλλάξει η κατάσταση αυτή στο μέλλον. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη έχει να κάνει με το Brexit. Το Λονδίνο μέχρι στιγμής αποτελούσε το οικονομικό κέντρο της Ευρώπης. Και της Ευρωζώνης βέβαια, έτσι δεν είναι, κατά κάποιο τρόπο. Αν αποχωρήσει λοιπόν τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος ήταν ο μελλοντικό ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Λονδίνο για την Ευρώπη των 27 ή για την Ευρωζώνη. Και πιστεύετε ενδεχομένω ότι διαδικασίες εκαθάρισης θα μπορούσαν να περάσουν στην Ευρωζώνη ή πιστεύετε ότι οι διαδικασίες αυτές θα παραμείνουν στο Λονδίνο με το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει αποχωρήσει όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εύκολα τα ερωτήματα αυτά. Λοιπόν, για ποιο λόγο είναι τόσο κατακαιρματισμένος ακόμα ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Κοιτάξτε, ο κατακαιρματισμός αυτός είναι αποτέλεσμα της κρίσης. Της κρίσης που είχαμε στο τραπεζικό τομέα και στην αντίδραση των εθνικών και υποπτικών αρχών απέναντι στην κρίση αυτή. Εν μέρη λοιπόν είναι ιδιωτικοί φορείς, ιδιωτικοί παράγοντες αυτοί οι οποίοι αποσύρθηκαν αν θέλετε και γίνανε πολύ πιο περιφερειακοί και μεμονωμένοι. Και από την άλλη βέβαια υπήρχαν και οι ρυθμιστές που τους λέγανε ότι θα πρέπει να έχουν μια πιο έντονη εποπτική προληπτική δραστηριότητα, να είναι πιο προσεκτικές οι τράπεζες στη λειτουργία τους και στις διασυνοριακές λειτουργίες τους. Στόχος πάντως της τραπεζική Ένωσης να δημιουργήσει κοινού και νέου κανόνες για όλη την τραπεζική αγορά. Μία εποπτική αρχή, ενιαίοι κανόνες για όλους και κατά αυτόν τον τρόπο οι τράπεζε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν εύρυθμα και διασυνοριακά. Ασχολούμεθα ακόμα με την εθνική διακριτική ευχέρεια και τις εναλλακτικέ εθνικές επιλογέ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα νομίζω ότι ήδη από πέρυσι είχε καταρτήσει ένα τεράστιο κατάλογο 160 περίπου διαφορετικών κανόνων και ρυθμίσεων που ισχύουν ακόμα σε εθνικό επίπεδο. Βαθμία βέβαια προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν κάπως τον κατάλογο αυτό. Κάποιοι εθνικοί κανόνες αναγκαστικά θα παραμείνουν, άλλοι πάλι όμως θα εναρμονιστούν ή κάποιες αρμοδιότητες ή κάποιοι κανόνες θα αποτελέσουν πλέον αντικείμενο διαχείρισης των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Είναι σε εξέλιξη πάντως ακόμα η όλη διαδικασία. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε και διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασυνοριακές εργασίες, δραστηριότητες η τεχνολογία θα μας βοηθήσει επίσης. Βλέπετε ότι υπάρχουν τράπεζες οι οποίες ηγούνται των τεχνολογικών εξελίξεων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, τεχνολογική καινοτομία στις τράπεζες, το λεγόμενο FinTech, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όλο και περισσότερο και καταφέρνουν οι τράπεζες να προωθήσουν την χρηματοπιστωτική αυτή τεχνολογία με χαμηλό κόστος. Όσον αφορά τώρα το Brexit και το ρόλο του City του Λονδίνου. Προφανώς το City του Λονδίνου είναι το χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ευρώπης και νομίζω ότι θα παραμείνει ένα από τα σημαντικά χρηματοπιστωτικά κέντρα του κόσμου. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να καταρρεύσει το City του Λονδίνου και ότι όλοι θα αρχίσουν να τρέχουν μακριά από αυτό και να φεύγουν. Νομίζω ότι δραστηριότητες πρόσβασης στην αγορά και δραστηριότητες ρύθμισης ενδεχομένως να φύγουν από το Λονδίνο αλλά όχι στον βαθμό που ορισμένοι λένε όσον αφορά τις διαδικασίες εκαθάρισης από πλευράς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα ήταν χρήσιμο αν οι διαδικασίες αυτές ήταν λιγότερο συγκεντρωμένες και είχαν καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας δηλαδή. Και η διαδικασία αυτή εν ευθέτω χρόνο βέβαια θα λάβει χώρα, αλλά βέβαια αν οι δραστηριότητε αυτέ αρχίσουν να είναι ε, μοιρασμένε σε διαφορετικέ αγορέ και να εμφανίζονται σε διαφορετικέ χώρε και αγορέ, το κόστο αναγκαστικά θα αυξηθεί. Και πολλοί ανησυχούν γι' αυτό. Διότι χρησιμοποιούν αυτέ τι διαδικασίε εκαθάριση και προφανώ θέλουν να τι χρησιμοποιούν με το χαμηλότερο δυνατό κόστο. Ενδεχομένω λοιπόν να πρέπει να καταβληθεί ένα τίμημα όσον αφορά την ε, μελλοντική διευθέτηση αυτών των δραστηριοτήτων. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Παδημούλης έχει το λόγο. Κύριε Ντάισελμπλουμ, σας καλωσορίζω για τελευταία φορά στην Επιτροπή μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι η πολιτική μου ομάδα και εγώ προσωπικά έχουμε συχνά διαφωνήσει και με την πολιτική που εκφράσατε τα προηγούμενα χρόνια ως πρόεδρος του Eurogroup και με ορισμένες δηλώσεις σας. Όσο όμως πλησιάζετε προς το τέλος της θητείας σας, και πιο πολλά καλά νέα μας φέρνετε και κάποιες αλήθειες μας τις λέτε και πιο ανοιχτά. Θα προτιμούσα αυτά να μας τα λέγατε και όταν ήσασταν πολύ ισχυρός πρόεδρος του Eurogroup. Όπως την αλήθεια ότι με το μνημόνιο και τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν για την Ελλάδα κυρίως σώθηκαν οι τράπεζες και όχι οι Έλληνες πολίτες όπως και με την αλήθεια που σήμερα μόλις είπατε ότι ο ελληνικός λαός που έχει υποφέρει πολλά από τα μνημόνια πληρώνει δύο πράγματα. Το πρώτο, την κακή διακυβέρνηση της πατρίδας μου για χρόνια από κυβερνήσεις που δημιούργησαν ελλείμματα και χρέη αλλά και τον κακό σχεδιασμό των προγραμμάτων. Σήμερα όμως, ακόμη και εσείς που είστε πολύ αυστηρός, μας είπατε πολύ καλά νέα ε, ε, για την Ελλάδα. Και εγώ θέλω σε αυτά να στηριχτούμε για να οικοδομήσουμε μια χώρα με ισχυρή διοίκηση, με μεταρρυθμίσεις, με ισχυρό κοινωνικό κράτος που να έχει βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό σας ρωτώ το εξής. Επειδή από το χρέος των 86 δισεκατομμυρίων ευρώ, από το δάνειο των 86 δισεκατομμυρίων ευρώ του τρίτου προγράμματος, ε, ο κύριος ε, Ρέκλινγκ έχει πει ότι ένα μέρος που δεν χρησιμοποιήθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα μπορούσε να δοθεί για την εξόφληση δανείων προς το IMF για παράδειγμα που έχουν υψηλά επιτόκια. Εσείς προσωπικά υποστηρίζετε αυτή την πρόταση ως ένα συγκεκριμένο μέτρο ελάφρυσης του ελληνικού δημόσιου χρέους που δεν θα δημιουργούσε πρόσθετο βάρος για κανέναν. Και δεύτερον, έρχεστε συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως το Eurogroup δεν έχει καμία υποχρέωση λογοδοσίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την άποψη να είναι υποχρεωμένο το Eurogroup να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια θεσμική αλλαγή. Πώς τη βλέπετε. Και τελευταίο, θέλω ένα σχόλιο, μια αξιολόγηση δική σας για το διάδοχό σας τον κύριο Σεντένο καθώς ήταν για καιρό μέλος του Eurogroup. Thank you. There are actually some obligation and this, meeting is... Υπάρχουν κάποιες ε, υποχρεώσεις. Η συζήτηση βέβαια είναι ανοιχτή. Ε, thank Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδημούλη. Πράγματι, έχετε παρακολουθήσει πολύ επικριτικά τη δουλειά που κάναμε και εντάξει αυτό δεν είναι μόνο η δουλειά σας και η υποχρεωσή σας αλλά ε, ιδιαίτερα επίμονοι στην επικριτική σας, στην κριτική σας. Ε, έχω συχνά πει ότι οι Έλληνε πολιτικοί είναι τόσο επικριτικοί για τι αποφάσει του παρελθόντο όσο ήμασταν και εμεί για τα λάθη που κάναμε στι αρχέ τη κρίση, όπω μόλι ανέφερα ε, και αυτό μπορεί να μα βοηθήσει ώστε να βελτιωνόμαστε για το μέλλον. Ε. Για το ερώτηση, την ερώτησή σας για την ε, ε, πρόορη πληρωμή των δανείων του Δουνουτού, αυτή ήταν η ερώτησή σας. Ναι, υπάρχει επιθυμία στο Eurogroup να παραμείνει το IMF σε αυτό το πρόγραμμα. Και όντως επί της αρχής έχει συμφωνήσει να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά ακόμα δεν έχει βάλει τη λεφτά. Μάλλον, συγγνώμη, δεν έχει... Ε, ε, δεν το έχει κάνει πράξη και υποτίθεται θα ξεκινήσει από την αρχή του επόμενου έτους. Ταυτόχρονα το να ξεπληρωθούν τα δάνεια του Δουνουτού ε, πράγμα που θα το κάνει να, να είναι λιγότερο αναμειγμένο. Ενώ ακόμα συζητάμε τη συμμετοχή και σε αυτό το πρόβλημα. Ναι, είναι λίγο σόλικο. Από οικονομική άποψη το καταλαβαίνω. Γιατί τα δάνεια του Δουνουτού είναι πιο ακριβά, ενώ τα ευρωπαϊκά είναι πιο φθηνά. Όταν μιλάμε για θέματα χρέους, τα οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν πολύ αργότερα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και αν ολοκληρωθεί επιτυχώς τόσο το καλύτερο. Θα δούμε την βιωσιμότητα του χρέους και για τα και πιο μακροπρόθεσμα στο να δούμε τι ακόμα πρέπει να γίνει. Εάν θέλουμε να μειώσουμε το βάρος του χρέους, είναι μια από τις δυνατότητες αυτή να αλλάξουμε το πακέτο των, των δανείων. Αλλά υπάρχει από την άλλη πλευρά το πολιτικό ζήτημα ότι θέλουμε να παραμείνει το ΔΝΤ και να παραμείνει υπεύθυνο και αυτό για το ελληνικό πρόγραμμα. Οπότε οριστική απάντηση δεν μπορώ να σας δώσω, εξαρτάται από το Eurogroup. Το Eurogroup ε, υπόλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε κάνει συχνά αυτή τη συζήτηση. Εγώ εκτιμώ την κοινοτική μέθοδο, αλλά δεν χρειάζεται να αποκλεί τη διακυβερνητική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Εάν θέλουμε να προοδεύσουμε στην Ευρώπη και αυτό που κάνουμε να τα κάνουμε πιο ισχυρά, μάλλον θα πρέπει να είναι ένα συνδυασμό. Κάποιε φορέ κοινοτική μέθοδο, κάποιε διακυβερνητική. Το γεγονό ότι εγώ είμαι εδώ σήμερα, ας πούμε, είναι μια σύνδεση ανάμεσα στη διακυβερνητική ομάδα των Υπουργών και το ίδιο θα ισχύσει και, και το Κοινοβούλιο. Και ε, δεν μπορεί να είναι πάντα όλες οι χώρες και αυτό πρέπει να το δεχτούμε. Και το Eurogroup είναι ένα παράδειγμα αυτού, γιατί είναι μια επιλογή σημαντική και ευρεία των ευρωπαϊκών χωρών που αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτό το project, θα συνεχίσουν. Δεν είναι όλοι και οι, 10, και οι 27. Ίσως στο μέλλον. Αλλά αυτό δεν θα μας σταματήσει για την ώρα. Οι δύο μέθοδοι λοιπόν, κοινοτική και διακυβερνητική, θα συνεχίσουν να ε, συνεπάρχουν. Και βεβαίως θα υπάρχουν και τριβές ανάμεσα στις δύο. Τέλος. Για τον συνάδελφο Μάριο Σεντένο είμαι πολύ ευτυχής για αυτή την επιλογή και τον ε, συνεχάρην και εδώ ε, για την ανάληψη των νέων αυτών αρμοδιοτήτων. Πιστεύω πως η επιτυχία της Πορτογαλίας που κατάφερε να βγει από το πρόγραμμα σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και, ε, οφείλεται και στην προηγούμενη κυβέρνηση γιατί έλαβε πολύ δύσκολες αποφάσεις όμως η Πορτογαλία τα πάει πάρα πολύ καλά ο Μάριο Σεντένο το έχει αυτό διαχειριστεί πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και είναι μια συμβολική ανταμοιβή για τις προσπάθειες που κατέβαλε το γεγονό ότι είναι τώρα ή μάλλον θα αναλάβει τον Ιανουάριο την Προεδρία του Eurogroup και εύχομαι κάθε επιτυχία. Thank you. Uh, Sven Σε ευχαριστώ, Σβέν Γκίγκολ. Θα μιλήσω γερμανικά για να εκφραστώ με ακρίβεια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εξ ονόματος της ομάδας μας για τη συνεργασία και εύχομαι καλή συνέχεια και ελπίζω να συνεχίσετε να υπηρετείτε τα δημόσια πράγματα. Ε, επιπλέον, εκτιμούμε την συνεισφορά σας, ε, ας πούμε, σε δύσκολους ε, καιρούς που έπρεπε να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις για την Ελλάδα και καταφέρατε να υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup, κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο και καταφέρατε να διατηρήσετε την ενότητα σε δύσκολες στιγμές. Ε, επί σειρά ετών είχαμε τις διαφωνίες μας, ε, ειδικά για θέματα φορολογικά, ειδικά στη δική σας χώρα θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα πράγματα. Ε, για το θέμα γενικά της πλευράς των εσόδων και των δαπανών, αλλά τελικά το ερώτημα που προκύπτει στο τέλος της εντολής σας είναι ο θεσμικός ρόλος του Eurogroup. Ξεκινήσατε κάποιες ε, μεταρρυθμίσεις τις οποίες ε, χαιρετίζουμε για περισσότερη διαφάνεια αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει ότι λαμβάνει το Eurogroup αποφάσεις ε, για μεταρρυθμίσεις οι οποίες εντάξει δεν εφαρμόζονται, βυθίζουν εκατομμύρια ανθρώπους στην ε, ανεργία, οι αποφάσεις αυτές, ε, αλλά ποιος φέρει ποιο μέρος της ευθύνης σε αυτές τις αποφάσεις, ποιος είχε ποια θέση, μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό, δεν υπάρχει διαφάνεια. Έτσι δημιουργείται ένα κενό λογοδοσίας. Αυτό το κενό λογοδοσίας δεν μπορεί να καλυφθεί. Και γνωρίζουμε σήμερα για διαφωνίες όπου οι ή και αντιφάσεις όπου οι υπουργοί εντό του Eurogroup λέγαν άλλα πράγματα από ό,τι λέγαν μετά όταν βγαίνανε στα ΜΜΕ και στη Γερμανική Βουλή και στο κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο. Ε, λοιπόν να είναι ανοιχτό το ερώτημα προς σας και αυτό το οποίο μπορείτε να συνεισφέρετε για τη λογοδοσία και τη δημοκρατία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι πρόσβαση περισσότερη στα έγγραφα, τουλάχιστον τα έγγραφα και τα πρακτικά αν υπάρχουν των Eurogroup των τελευταίων ετών να γίνουν δημόσια έτσι ώστε να μπορούν να οδηγηθούν και στην κάλπη οι πολίτες έχοντας γνώση των ε, πραγμάτων. Τουλάχιστον λοιπόν, έστω με κάποια χρονική καθυστέρηση, θα πρέπει να μαθαίνουν και να πληροφορούνται οι πολίτες ποιος υπουργό είχε ποια τοποθέτηση και ποια θέση. Νομίζω ότι μέχρι τον Ιανουάριο μπορείτε κάτι να κάνετε, κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα ε, ήταν ε, υπέρ σας και στον τελικό απολογισμό της ε, θητείας σας. Ευχαριστώ κύριε Γκίγκολτ. Είπατε κάποια πράγματα φιλικά, κάποια άλλα. Όχι και τόσο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια λοιπόν. Είπατε ότι ήμουν κάπως πιο ήπιος μαλθακός στην πλευρά των φόρων. Ε, είναι ευαίσθητο αυτό το θέμα γιατί διαφωνώ ριζικά. Είπα και πριν ότι η φορολογική πολιτική της Ολλανδίας ε, δεν βοηθάει ε, προσθέτει στο πρόβλημα και ότι πρέπει να γίνουμε μέρος της λύσης. Και τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουμε αλλάξει τελείως στρατηγική. Μπορεί να μην το αναγνωρίζετε, να μην θέλετε να το αναγνωρίσετε δημοσίω, αλλά είναι αλήθεια. Έχω καταβάλει μεγάλες προσπάθειες κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας ε, το 2016 σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για την οδηγία φοροαποφυγής, κατά της φοροαποφυγής που περιείχε 5-6 προτάσεις και πριν το τέλος του έτου είχαμε συμφωνία και για την δεύτερη σχετική οδηγία που ήταν πολύ ακαθόδε θέμα στην Ολλανδία γιατί ακριβώς έπλητε μια δομή που είναι πολύ σημαντική για τις αμερικανικέ εταιρείε που χρησιμοποιούσαν το Ολλανδικό φορολογικό σύστημα. Θεωρώ λοιπόν και οπωσδήποτε και η δική σας η πίεση και η πίεση του Κοινοβουλίου βοηθούσε ε, στο να σημειώσουμε σοβαρή πρόοδο τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Αυτά. Ε, Βεβαίω ποτέ δεν ε, ολοκληρώνεται αυτή η δουλειά και πρέπει να συνεχιστεί. Για την διαφάνεια. Προσπάθησα να την βελτιώσω δεδομένου του ότι είναι ένα διακυβερνητικό πλαίσιο και είναι άτυπες οι συναντήσεις Ε, έτσι είναι το, το Eurogroup. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έκανα ό,τι μπορούσα για να βελτιώσω την διαφάνεια όλα τα έγγραφα ακόμα και άλλων θεσμικών οργάνων, οτιδήποτε υπήρχε, πιέσαμε για να δημοσιεύονται πριν την ε, συνεδρίαση, οπότε και ο εξωκόσμος πληροφορείται το τι θα συζητήσουμε ε, κάνω ό,τι μπορώ στην πλευρά της επικοινωνίας ε, και πολλά έχω δημοσιεύσει ε, συχνά μετά τις συναντήσεις. Όταν μιλάτε λοιπόν για πρακτικά και έγγραφα αυτά έχουν ήδη γίνει. μιλάτε επίσης για παρελθόντα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Αυτό είναι πάντα δύσκολο γιατί θα έπρεπε οι Υπουργοί εκ των προτέρων να γνωρίζουν ότι θα δημοσιοποιηθούν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο. Και για να γίνει αυτό εκ των υστέρων δεν μου φαίνεται σωστό. Τέλος πάντων, πότε ελήθησαν αυτές οι αποφάσεις το, το 16. Ε, έκτοτε λοιπόν όλα τα έγγραφα που συντάσσονται για το Eurogroup και για τους υπουργούς και η ημερήσια διάταξη με τις ε, σημειώσεις. Όλα αυτά δημοσιεύονται όπως ε, και τα πρακτικά εκ των υστέρων. Αυτά. Νομίζω έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο σε αυτό. Μα έχουν δημοσιευτεί και τα πρακτικά των ε, ε, Υπουργικών ε, Συμβουλίων του Πολέμου. Ελπίζω να μην χρειάζεται να περιμένουμε τόσο. Ε, αυτά είναι οι κανόνες των εθνικών αρχείων, λέει ο πρόεδρος. Μία παρατήρηση, γιατί θυμάμαι μία συζήτηση που είχαμε μετά την απόφαση για την Κύπρο. Ο κύριος Γκίγκολτ ζητούσε ποιος έλαβε ποια απόφαση εντός της αιθούσης του Eurogroup. Και έλεγα τότε και θα συνεχίσω να λέω ότι ήταν μία κοινή απόφαση που λήφθη ομόφωνα και αν κάποιος συνάδελφος στο κοινοβούλιο του είπε κάτι το διαφορετικό, όπως ε, υπονοήσατε, τότε ε, ίσως δεν ήταν ειλικρινής. Ήταν μια κοινή, ομόφωνη απόφαση και, επί το αποτέλεσμα για την ε, Κύπρο και το κυπριακό πρόγραμμα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό από ότι το πρόγραμμα για την Ελλάδα. Και αυτό έχει σχέση με τη διαφορετική προσέγγιση που είχαμε στην Κύπρο, για το οποίο μου ασκήθηκε κριτική ξανά και ξανά και πράγμα το οποίο θα υπερασπίζομαι ξανά και ξανά. Και το αποφάσαν όλοι οι παρόντες υπουργοί. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άνεμαντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει η εντύπωση από την ε, συζήτηση ότι δεν θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα για το πώς βλέπετε το μέλλον της Ευρωζώνης γιατί εγώ θα επιμείνω όμως γιατί εντάξει ο ρόλος σας ε, είναι κάπως ε, συμβολικός. Ναι βεβαίως ο διάδοχός σας πρέπει να ανταμυφθεί για την πολιτική που ακολούθησε η Πορτογαλία, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα ε, από ένα σοσιαλιστικό κόμμα το οποίο είναι κατά οποιασδήποτε πολιτικής ε, συγκράτησης των δημοσίων δαπανών και από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με κάποιο έγγραφο της ε, Κομισιόν φαίνεται πως αρκετές χώρες φοβόντουσαν για την σταθερότητα και την ανάπτυξη της Ισπανίας και άλλων χωρών. Οπότε το ερώτημά μου είναι αν συμφωνείτε ότι η αποχώρησή σας είναι σύμβολο για το τέλος της πολιτικής ε, λιτότητας ε, και για μια αλλαγή ε, πολιτικής κατεύθυνσης. Και αν δεν συμφωνείτε να μου πείτε γιατί. Σας ευχαριστώ κύριε Χάναμανς ε, για την ερώτησή σας. Χαίρομαι για την ερώτηση. Είναι ενδιαφέρουσα ε, και η συζήτηση που γίνεται στα ΜΜΕ για το εάν η πορτογαλική κυβέρνηση στηρίζει την δημοσιονομική πολιτική, ή την απορρίπτει και το τι σημαίνει αυτό για την πολιτική της Ευρωζώνης. Πρώτα απ' όλα η στρατηγική του Eurogroup ποτέ δεν ήταν λιτότητα τελεία. Αυτή είναι η ρητορική και αυτή είναι η συζήτηση που ε, γίνεται, αλλά η στρατηγική πάντα αφορούσε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, το να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, πιο ανθεκτικές οι οικονομίες, να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Δεύτερον, πιο βιώσιμα δημόσια οικονομικά. Σταδιακά βεβαίω. Είναι μια αργή διαδικασία. δεν έχει ολοκληρωθεί σε αρκετές χώρες, οπότε η στρατηγική πάντα ήταν δυτή και προς τρεις ε, κατευθύνσεις. Δεν ήταν μόνο θέμα ε, ισοσκελισμού του προϋπολογισμού. Αυτό είναι παρεξήγηση. Η Πορτογαλία ως ε, ένα έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στι δημοσιονομικές πολιτικέ και η κυβέρνηση δεν έχει αποκλίνει από αυτήν την πορεία. Και ο Πορτογάλος συνάλφος ήταν σαφές ότι η Πορτογαλία θα πρέπει να συνεχίσει σε αυτήν την πορεία προς τα βιώσιμα δημόσια οικονομικά δηλαδή. Οπότε αν η ερώτηση είναι εάν ε, ο νέος Υπουργός Πορτογάλος είναι κατά της λιτότητας. Αυτό είναι συζήτηση χωρίς αντικείμενο. Η στρατηγική του Eurogroup δεν είχε ποτέ οριστεί ε, από μια μονοδιάστατη προσέγγιση ποτέ ως λιτότητα. Οπότε η στρατηγική μας δεν θα αλλάξει ουσιαστικά. Μεγάλο κομμάτι της στρατηγικής βεβαίως ε, είναι ενσωματωμένο στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τις άλλες ε, συμφωνίες που έχουμε. Ένα άλλο κομμάτι είναι το να ξεσκαρτάρει ο χρηματοπιστωτικός τομέας ε, και να ξαναρχίσει να λειτουργεί. Οπότε η αλλαγή της Προεδρίας δεν σημαίνει ότι ε, θα αλλάξουν οι πολιτικές. Έχουν καθοριστεί στις μεταξύ μας συμφωνίες και θα λαμβάνονται αποφάσεις τουλάχιστον στο Eurogroup ομοφόνος. Σας ευχαριστώ. Εστέρ Ντελάνγκε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στον πρώτο κύκλο μιλητών ακούσαμε διάφορα επίπεδα εκτίμησης ή απουσία εκτίμησης προς το έργο του Προέδρου του Eurogroup. Γενικά όμως ήταν θετικά τα σχόλια ενδεχομένως ε, πιο θετικά ακόμα και από πολιτικές ομάδες που δεν είναι καν στη δική σας την πολιτική οικογένεια. Αυτό μάλλον τι σημαίνει, ότι κάνετε μάλλον καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Όσον αφορά τι παρατηρήσει για Τραπεζική Ένωση, επ' αυτών θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτό το οποίο είπατε για τι πρόσφατε περιπτώσει εξυγίανση τραπεζών και πώ θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτή την εμπειρία όσον αφορά την ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση. Οι περιπτώσει όμω αυτέ εξυγίανση έδειξαν ότι οι εθνικέ θέσει αφετηρία, δηλαδή τα εθνικά πλαίσια, είναι αρκετά διαφορετικά αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήγεται δηλαδή στο συμπέρασμα ότι και για την ολοκλήρωση του τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης θα πρέπει να έχουμε μία κάποια δομή που να αφήνει μία κάποια ευθύνη μια κάποια αρμοδιότητα και για δημοσιονομικά θέματα ως προς το 0,8% των καλυμμένων καταθέσεων σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία δηλαδή με τα όσα αποφασίζονται για το ευρωπαϊκό επίπεδο Νομίζω ότι λόγω της μεγάλης αυτής διαφοράς που υπάρχει αυτή τη στιγμή από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, χρειαζόμαστε και αυτές τις εθνικές αρχές και σε εθνικό επίπεδο, να μπορούμε δηλαδή να τηρήσουμε και εκεί κάποιες ε, αρμοδιότητες για να αντιμετωπίσουμε μια ενδεχόμενη μελλοντική κρίση. Δεύτερη ερώτηση σε σχέση με τις παρατηρήσεις που κάνατε για το πώς ε, οι δέσμοι μέτρων για την Τραπεζική Ένωση και συγκεκριμένα μέτρα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια για άλλα προβληματικά ζητήματα θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρου πρόοδου. Είπατε ότι χρειαζόμαστε να σημειώσουμε πρόοδο και στη μείωση του κινδύνου και στον επιμερισμό του κινδύνου. Μόλον ότι μπορεί να με κατηγορήσει γι' αυτό η Περβόν Μπερέ, εγώ σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι θα έπρεπε να είχαμε ολοκληρώσει όλη την εργασία για τη μείωση του κινδύνου προτού προχωρήσουμε στην αμοιβαιότητα, στον επιμερισμό δεν θα πρέπει τουλάχιστον να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε μείωση του κινδύνου. Ποια στοιχεία θέλουμε να δούμε στα πλαίσια του μελλοντικού ευρωπαϊκού συστήματος διασφάλισης των καταθέσεων. Νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμα πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Επομένως, όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και ο πρόεδρο είπε ότι είναι θετικό να έχουμε, μάλλον ότι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμή είναι βίωνα. Ποιο όμως είναι το πλαίσιο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα επόμενα πέντε χρόνια, για παράδειγμα, προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε περισσότερο με τα δεδομένα τα οποία υφίστανται σε διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντελάνκη και ευχαριστώ και για τη στήριξή σας τα προηγούμενα χρόνια. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα ερωτήματά σας, οι περιπτώσεις εξυγίανσης. Κοιτάξτε, εδώ πέρα ακούσαμε διαφορετικές αντιδράσεις. Ορισμένοι είπαν ότι να, οι περιπτώσει αυτέ δείχνουν ότι απέτυχε η Τραπεζική Ένωση. Άλλοι πάλι είπαν ότι όχι, δείχνουν ότι λειτουργεί η Τραπεζική Ένωση. Εγώ νομίζω ότι καταδεικνύουν ότι λειτουργεί η Τραπεζική Ένωση, αλλά ότι απομένουν ακόμα κάποια κενά, κάποιε αδυναμίες τις οποίες θα πρέπει να καλύψουμε, πράγματα που δεν είχαμε καταφέρει να προβλέψουμε. Αυτό που είχαμε δει όμως εξ αρχής είναι ότι τα εθνικά συστήματα εξυγίανσης διαφέρουν πολύ το ένα από το άλλο ακόμα, όπως το είπατε κι εσείς. Και το ζήτημα γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκο, ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλά πολύπλοκα νομικά ζητήματα σε αυτά τα πλαίσια εξυγίανσης των τραπεζών σε εθνικό επίπεδο και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ιδίω όσον αφορά την εξυγίανση των τραπεζών. Αν ήταν κάποιο πολύ φιλόδοξο και θα αρελαίο, θα έλεγε ότι θα πρέπει να καταργήσουμε όλα αυτά τα εθνικά συστήματα και να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό ενιαίο μόνο σύστημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το πολύ δύσκολο που θα έχει και έντονες πολιτικές συνέπειες. Ανταυτού θα μπορούσαμε πέρα από το εθνικό επίπεδο και τα εθνικά πλαίσια εξυγίανσης να έχουμε και ένα ευρωπαϊκό επίπεδο εναρμονισμένο, όπου να μπορούμε τουλάχιστον για τον τομέα των τραπεζών να κινούμεθα πιο συλλογικά, πιο ενοποιημένα. Και θα πρέπει να δούμε έπειτα πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε τα πλαίσια αφαιρεκιότητας και τα πλαίσια εξυγίανση των τραπεζών. Δεν θα πρέπει να καταλήγουμε στα συστήματα αφαιρεγγιότητα μόνο και μόνο επειδή φαντάζουν να είναι πιο εύκολα, ενώ θα έπρεπε για ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για παράδειγμα, να ακολουθηθεί περισσότερο δρόμο τη εξυγίανση. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσπαθήσει όχι μόνο να ολοκληρώσει η Τραπεζική Ένωση, αλλά να δημιουργήσει και μία ένωση κεφαλαγορών. Να μπορούμε να έχουμε δηλαδή ένα πλαίσιο αφαιρεγγιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να βγει δηλαδή αυτό από το εθνικό επίπεδο και να μπορεί να λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου η κυρία Μπερές, πάντως βλέπω ότι γνέφει προς διάφορες όμως κατευθύνσεις. Τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την αρμοδιότητα. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί και η Ένωση Κεφαλαγορών. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια ένωση αν υπάρχουν τόσες πολλές εθνικές διαφορές. Το δεύτερο ερώτημά σας, τι χρειάζεται για τη μείωση του κινδύνου. Το θετικό στοιχείο του δικού χάρτη για την Τραπεζική Ένωση που αποφασίσαμε το 2016 είναι ότι συγκεκριμενοποιούσαμε πλέον τι θα πρέπει να γίνει για τη μείωση του κινδύνου και τον περιορισμό του κινδύνου, αλλά δεν ήμασταν αρκετά ακριβής για το πότε θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Και ορισμένες χώρες που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα για τον επιμερισμό του κινδύνου, για την αμοιβαιότητα του κινδύνου, το χρησιμοποίησαν αυτό, υποφελήθηκαν της ασάφειας αυτής, λέγοντας ότι δεν έχει έρθει ακόμα το πλήρωμα του χρόνου ή ότι θα πρέπει να περιμένουμε κτλ. Έτσι λοιπόν τη Δευτέρα στο Eurogroup καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι στο επόμενο πλέον στάδιο, βάσει του εγγράφου που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από δικό μας αίτημα, όπου βλέπουμε όλο το έργο το οποίο έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμή. Βάσει λοιπόν του εγγράφου αυτού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε πλέον να συγκεκριμενοποιήσουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θέλουμε να δούμε και πότε θα πρέπει αυτά να λάβουν χώρα. Πολύ εύκολο να το λέει κανεί αυτό, δυσκολότερο στην πράξη. Πάντω είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε ήδη από τη στιγμή αυτή να μιλάμε για το ADs για αυτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασφάλισης των Καταθέσεων και θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι πλέον. Τι μας ικανοποιεί, πότε θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο μας επιτρέπει να περάσουμε στο επόμενο. Ευχαριστώ. θα πρέπει να δούμε ποια είναι η συμμετρία ανάμεσα στα δύο επίπεδα. Όπως είπατε είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση που θα συνεχίσουμε Κώστας Μαυρίδης. Even though I'm tempted to speak about EDIS, uh, given that this is the last chance we had to have in front of us Mr. Dijsselbloem, I would rather to concentrate... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσω καλύτερα για το θέμα της Κύπρου και είσαστε ο κατάλληλος άνθρωπος με την ευκαιρία. Κύριε Ντάισελμπλουμ, ε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις ε, μελλοντικές σας, στη μελλοντική σας σταδιοδρομία. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της Κύπρου, είπατε πριν ότι το θυμάστε πολύ καλά και θέλω να σας θυμίσω κάποια από τα γεγονότα. Μάρτιος 2013. Το bail-in ήταν αναπόφευκτο, υποτίθεται. Ε, με βάση κάποια σενάρια. Μετά από μια μακρά συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών στο, Eurogroup, ανακοινώθηκε η αποκαλούμενη πρώτη πρόταση Μπέιλιν συμπεριλαμβανομένων των ε, εξασφαλίσεων για τις ε, καταθέσεις. Μετά από την παρέμβαση της ΕΚΤ την επόμενη μέρα αυτό το λάθος διορθώθηκε ώστε δεν υπήρχε καμία κανένας φόρος στις ασφαλισμένες ε, καταθέσεις. Ο γρίφος είναι ο εξής. Αν και περιμέναμε να, γίνει, να υπάρξει bail-in οριζόντιο για όλες τις τράπεζες, τελικά καταλήξαμε με ένα το οποίο ήταν επικεντρωμένο σε δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου. Η μία έκλεισε και η άλλη ήταν περίπου 50% των bail-in των καταθέσεων πάνω και πέρα από τις ε, ασφαλισμένες καταθέσεις. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς ξεκινήσαμε με οριζόντια ζώδιο Μπέιλιν και καταλήξαμε σε ένα σενάριο όπου ε, εστιάστηκε σε δύο συστημικές τράπεζες ενώ το αναμενόμενο θα ήταν μια εκδοχή του οριζοντίου με εξαίρεση των ε, των ασφαλισμένων καταθέσεων. Επίση, γνωρίζετε ότι τώρα που μιλάμε οποιοδήποτε, ευρωπαϊο πολίτη από την Κύπρο δεν μπορεί να ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα στο Βέλγιο. Ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια σε σχέση με το μέλλον μου. Εσείς επανέρχεστε σε αποφάσεις που ελήφθησαν το αρχές του 2013. Πρώτα απ' όλα, νομίζω πως όλοι συνειδητοποιούμε ότι η κατάσταση στην Κύπρο είχε αφαιθεί ε, ανεξέλεγκτη. Το πρόγραμμα για την Κύπρο θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, ε, νομίζω γιατί υπήρχαν οι εκλογές και περιμέναμε. Α, όταν εγώ ανέλαβα το Φεβρουάριο του 2013, ότι δεν μπορούσαμε να το καθυστερήσουμε άλλο. Θα ήταν πολύ καλύτερο αν η κατάσταση είχε αντιμετωπιστεί νωρίτερα και αν το πρόγραμμα είχε ε, ξεκινήσει νωρίτερα. Έχετε δίκιο ότι υπήρξαν δύο αποφάσεις. πρώτα, υπήρχε πολύ έντονη αίσθηση στο Eurogroup ότι η προσέγγιση του Μπέιλιν ήταν ε, αναπόφευκτη από την αρχή. Η, Κυπριακή κυβέρνηση όμως δεν ήθελε αυτή την προσέγγιση γι' αυτό και καταλήξαμε σε αυτήν την προσέγγιση και μας είπατε ότι ε, και μάλλον ε, καταρχάς επιβάλαμε φόρο σε όλους τους ε, λογαριασμούς, σε όλες τις τράπεζες και για όλους. Ήταν φόρος αυτός, φόρος ε, συμβολή για να σωθεί το οικονομικό σύστημα της Κύπρου. Τώρα αν αυτό ήταν ε, δικαιολογημένο ή όχι, το θέμα κλειδί ήταν ότι εδώ το μέγεθος των καταθέσεων δεν υπήρχε πραγματικό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων στην Κύπρο καθόλου. Η ασφάλιση των καταθέσεων σε εκείνη τη φάση στην Κύπρο ήταν ε, μύθος και οι επικρίσεις που είχαμε ήταν ότι η ε, ε, ήταν επίσης μύθος γιατί η Κύπρος ποτέ δεν θα, μπορούσε, δεν θα είχε μπορέσει να σώσει όλες τις καταθέσεις που υπήρχαν στις τράπεζες. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και η, προσέγγιση Μπέιλιν δεν υποστηρίχθηκε από την Κυπριακή κυβέρνηση και γι' αυτό και επιβάλαμε αυτό το φόρο. Ε, για, ε, το, όχι εκτε, αλλά το Κυπριακό Κοινοβούλιο ήταν αυτό που απέρριψε τη λύση και επανήρθαμε στην αίθουσα και ξαναδιαπραγματευτήκαμε και επιλέξαμε τη λύση Μπέιλιν που προτίμησαν οι περισσότεροι υπουργοί και θεσμοί στο Eurogroup από την αρχή. Εγώ έτσι θυμάμαι να γίνανε τα πράγματα. Και η κυβέρνηση της Κύπρου συμφώνησε στη δεύτερη πρόταση. Ναι, βεβαίως, αλλιώς δεν θα είχαμε λάβει αυτή την απόφαση. Πρέπει να καταλάβετε ότι η αντίθετη προσέγγιση, αν είχε υπάρξει δηλαδή δηλαδή bail-out των τραπεζών και πλήρης προστασία όλων των επενδυτών, αυτό θα είχε χρεοκοπήσει την Κύπρο τελείως. Ε, το να επιλέξουμε την προσέγγιση του bail-in για την Κύπρο, στην ουσία μείωσε το τεράστια δαπάνη για την Κύπρο και γι' αυτό μπορέσαμε να, περιορίσαμε το, να περιορίσουμε το, project, το πρόγραμμα για, στα 10 ε, δις. Αν είχαμε βάλει όλες τις τράπεζες και τις μεγάλες τράπεζες που είχαν ε, αναδιαρθωθεί και τα λοιπά, αν τις είχαμε κάνει bailout, τώρα η Κύπρος θα είχε πολύ πολύ μεγαλύτερο χρέος. Και μέχρι και σήμερα είμαι πολύ ευτυχής που δεν ακολουθήσαμε αυτό τον δρόμο. Αυτή την προσέγγιση συζητήσαμε και για την Ελλάδα. Και για bailout των τραπεζών. Είναι πάρα πολύ δαπανηρό και άδικο. Ε, γι' αυτό η Ελλάδα έχει ακόμα τόσο μεγάλο χρέος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντάισεμπλουμ, σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ε, εσείς ε, μπορεί να καταλήξετε να πάρετε σύνταξη βεβαίως ε, οι άλλοι άνθρωποι όταν φτάνουν σε αυτό το σημείο κάνουν έναν απολογισμό με ένα ποτήρι κρασί, ένα καφέ λοιπόν πρώτα απ' όλα κάποια πράγματα για τον απολογισμό της μέχρι τώρα πορεία σας ε, μήπως θα ήταν ε, καλύτερα να έχουμε κάποια πιο ισχυρά μέσα όσον αφορά την, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και την εδραίωσή του στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το πώς έχει στηθεί η ΙΟΝΕ. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την κρίση και μετά το 2008 έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα στην Ευρωζώνη. Έχει γίνει κάπως ισχυρότερη νομισματική ένωση. Είπατε και εσείς ο ίδιος ότι τα πράγματα άλλαξαν, αλλά έχουν γίνει αρκετά τώρα για να πούμε ότι μπορούμε να αποφύγουμε ε, μια τέτοια κρίση αν συμβεί αύριο, τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κρίσης αν συμβεί αύριο ξανά το ίδιο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ που θέλετε να μου δώσετε από τώρα σύνταξη. <laughs> Θα δω αν θα ζητήσω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είμαι πολύ νέος ακόμα, εν πάση περιπτώσει δεν θα γίνει αυτό. Τώρα για την εφαρμογή των ε, συγκεκριμένων συστάσεων αναχώρα ε, ήταν η εφαρμογή της πράγματι πολύ ασθενής και όμως αν δείτε τις εκθέσεις του ΩΣΑ για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν σε ολόκληρη την Ευρωζώνη είναι πολύ εντυπωσιακή. Βεβαίω, εντάξει δεν είναι αναχώρα. Κάποιες χώρες έχουν κάνει πολύ λίγα. Άλλες χώρες αναγκάστηκαν από τι περιστάσεις ή από προγράμματα να κάνουν πολύ δύσκολες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ενδιαφέρον είναι ότι αν δείτε την Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή οι χώρες με την υψηλότερη ανάπτυξη είναι οι χώρες οι οποίες έκαναν τις δύσκολες διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις τα προηγούμενα χρόνια. Η Ιρλανδία βεβαίως, η Πορτογαλία, οι Βαλτικές ε, χώρες ε, και η Ολλανδία θα έλεγα δείχνουν σημάδια πολύ ισχυρή ανάπτυξης μετά από την λήψη δύσκολων μέτρων. Τώρα, αν θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εφαρμογής ε, ή επιβολής ε, των συστάσεων αναχώρα. Προσωπικά, αν δείτε πόσο πολιτικό αγώνα δίνουμε για την εφαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου, φαντίζεστε τον πόλεμο που θα ξεσπάσει εάν η Κομισιόν πραγματικά παρεμβαίνει και λέει τώρα πρέπει να προσαρμόσετε την αγορά εργασία να κάνετε βιώσιμο το συνταξιδοτικό κτλ. Οπότε νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα του να αγκαλιάζει κάθε χώρα το, το πρόγραμμα. Η Κομισιόν λέει επίσης ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο μακροπρόθεσμα σε μια πολυετή προσέγγιση και να συμφωνούμε με την κυβέρνηση τι θα κάνετε τα επόμενα τρία χρόνια ως μεταρρυθμίσεις και βεβαίως τάξη, μπορεί να ασκήσει κριτική η Κομισιόν και να πει αυτό δεν αρκεί, πρέπει να αντιμετωπίσετε το χ και το ψ. Να υπάρχει δηλαδή μια τριετής συμφωνία και ίσως να συνδεθεί αυτό, αν απαιτείται, με κάποια στήριξη των μεταρρυθμίσεων και ίσως έχει η κομισιόν κάποια σχετική πρόταση για να στηρίξει χώρες οι οποίες κάνουν μεταρρυθμιστικές προτάσεις. Ε, μια πιο πολυετή προσέγγιση λοιπόν, όπου τα κράτη-μέλη παίζουν τον ηγετικό ρόλο, αυτά προτείνουν το τι θεωρούν ότι πρέπει να γίνει τα επόμενα τρία χρόνια και μετά από διάλογο με την Κομισιόν καταλήγουν σε κάποια συμφωνία. Νομίζω αυτό θα είναι πιο πολύτιμο από αυτό το οποίο γίνεται τώρα, ότι Κάθε χρόνο δηλαδή η Κομισιόν λέει αυτέ είναι οι συστάσει ένα χώρο, αυτό πρέπει να κάνετε και οι κυβερνήσει λένε ναι, αλλά εγώ σχεδιάζω να κάνω κάτι άλλο. Το θέμα είναι λοιπόν να τα αγκαλιάσουν αυτά τα κράτη-μέλη. Τώρα, αν έχω εμπιστοσύνη, αν ξεσπούσε νέα κρίση. Όχι, όχι ακόμα. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί είναι θέμα αντοχής ε, στους ε, κραδασμούς που μπορούμε να απορροφήσουμε Κάποιε Κάποιες χώρες εξακολουθούν να έχουν πολύ μικρό δημοσιονομικό περιθώριο για να αντιδράσουν σε οικονομικούς κραδισμούς μέσω μια πιο εκτατική ε, δημοσιονομικής πολιτικής. Δηλαδή, για κάποιες χώρε είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Οι τράπεζες μας ε, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά όχι όλε ακόμα και θα έλεγα ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης ε, κραδασμών, ε, περισσότερα αποθέματα, περισσότερο κεφάλαιο και πιο υγιείς ισολογισμούς ε, και νομίζω έχουμε βελτιωθεί και τα νοικοκυριά επίσης είναι πολύ ευπαθή ακόμα. Το ιδιωτικό χρέος σε κάποιες χώρες είναι πολύ υψηλό και αν υπάρξει κάποιο σοκ ε, θα είναι δύσκολα τα πράγματα εάν ε, καταρρεύσουν παραδείγματος χάρη οι αγορές ε, των ακινήτων και έχει κάποιος και έχουμε μεγάλο ποσοστό στεγαστικών βεβαίως υπάρχει πρόβλημα οπότε αν η περίοδος αυτής ανάπτυξης είναι μεγάλη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο για να δημιουργηθεί κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο για να δημιουργηθούν αποθέματα σε επίπεδα εταιριών, τραπεζών, νοικοκυριών και κρατών. Πρέπει να γίνουμε πιο ανθεκτικοί στις ε, αναταράξεις. Αλλά αυτό είναι αμυντική προσέγγιση. Θα πρέπει να έχουμε και μια επιθετική προσέγγιση, να φροντίσουμε να συνεχιστεί η ανάπτυξη, να γίνουμε ανταγωνιστικοί, να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας, να έχουμε καινοτομία στην Ευρώπη κτλ. Υπάρχει λοιπόν η άμυνα, θα έλεγα, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης κρασμών και η επίθεση, να γίνουμε πιο ε, δυνατοί. Και πρέπει να γίνει δουλειά και στα δύο μέτωπα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε Σίλβα Περίρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω πορτογαλικά. Μόλις αυτές το Eurogroup εξέλεξε ένα νέο ε, πρόεδρο, τον ε, Υπουργό Οικονομικών της Πορτογαλίας, τον ε, κύριο Σεντένο. καλός ιονός για το μέλλον του Eurogroup αλλά και για την Πορτογαλία Νομίζω ότι ο κύριος Ντάσελ σωστά υπογράμμισε την πρόοδο που έκανε η Πορτογαλία τα τελευταία χρόνια, καθώς επίσης ε, χάρη στην εξαιρετική του μνήμη θα θυμάται βέβαια ότι Ακόμα πριν από ένα χρόνο συζητούσαμε κυρώσεις κατά της Πορτογαλίας γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επιδεινώσει το διορθωτικό χρέος. Πολλά πράγματα άλλαξαν, η πορτογαλική οικονομία αναπτύσσεται, το χρέος μειώνεται, η Πορτογαλία βγήκε από τη διαδικασία υπερβολικού χρέους και η βαθμολογία της χώρας μου ε, βελτιώνεται και ο Υπουργός Οικονομίας μας είναι πρόεδρος τώρα του Eurogroup. Οι πολιτικέ ε, θα αλλάξουν ή δεν θα αλλάξουν στο μέλλον, δεν το ξέρουμε ακόμα. Όμω, ο Ντάισερ μου ξέρει όπω κανεί άλλο στο Eurogroup και θα ήθελα τη γνώμη σα ε, για τι προπτικές ε, με την πολιτικό, το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στο Eurogroup για ένα από τα βασικά προβλήματα του ενιαίου νομίσματο που είναι η απόκληση των οικονομιών. Πώ μπορεί αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί και εδώ τίθεται τα εξή. Σε ποιο βαθμό η νέα δημοσιονομική δυνατότητα ότι της Ευρωζώνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να καταπολεμηθεί η απόκληση αυτή και κατά δεύτερο λόγο πώς γίνεται να είναι δυνατόν να καταπολεμηθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες με τη μορφή των ε, δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Εσείς είπατε σήμερα ότι είναι σημαντικό οι χώρες με δημοσιονομικό περιθώριο να επενδύουν περισσότερο για να προωθήσουν την ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα μήνυμα θετικό, αλλά τα μέσα είναι αδύναμα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύω πως μια μεταρρύθμιση τη Ευρωζώνης θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία πιο, πιο συμπαγών και στεναρών εργαλείων, ώστε οι χώρε που έχουν περισσότερο όντω περιθώριο δημοσιονομικό να κάνουν περισσότερε επενδύσεις για να περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Um, so, uh, thank you, uh, Silva Pereira, for your questions. Ευχαριστώ κύριε Σίλβα Περέιρο για τις ερωτήσεις σας. Κάνατε μια παρατήρηση για την προηγούμενη κυβέρνηση της Πορτογαλίας και ως πρόεδρος του Eurogroup έχω συνεργαστεί πολύ στενά και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Θα πρέπει να πούμε και τα καλά, έκαναν δύσκολη και σημαντική δουλειά για να βγει η Πορτογαλία από την κρίση. Δεν είναι δίκαιο να μην το πούμε. Εγώ εργάστηκα πολύ στενά με τη Μαρία Λουίζα Αλμπουκερούγη, πολύ καλή υπουργό οικονομίας και πολύ ε, ξεσέβαστη στο Eurogroup. Υπάρχουν ε, αποκλήσεις ναι, ανάμεσα στην οικονομική και δημοσιονομική θέση της κάθε χώρας, στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι πολιτικός περίπλοκο και είναι δύσκολο να το χειριστούμε, να έχουμε αποτελεσματικές ε, ε, πολιτικές, γιατί αν ήμασταν όλοι στην ίδια φάση του κύκλου θα ήταν πολύ πιο εύκολο να σχεδιάσουμε την οικονομισματική πολιτική για όλους. Όμως οι διαφορές υπάρχουν. Ε, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος σε χώρες που βρίσκονται ήδη στο πάνω μέρος του κύκλου ε, και έχουν πλήρη απασχόληση και θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερο και να σπρώξουν ακόμα περισσότερο την οικονομία τους και να δημιουργήσουν ενδεχομένω φούσκες ενώ σε άλλες χώρες θέλουμε περισσότερες επενδύσεις σε δημόσιες. Είναι πολύ θέμα κλειδί αυτό βέβαια, αλλά δείχνει επίσης ότι τη βασική ευθύνη για τη δημιουργία περισσότερο ισορροπημένης θέσης ε, τη φέρει το εθνικό επίπεδο. Συχνά λέω ότι τα κρατη και η εθνική πολιτική ε, εξαιρετικά συχνά κατηγορούν την Ευρώπη και την Ευρωζώνη για τα προβλήματά τους ε, και πολύ συχνά επίσης περιμένουν λύσεις για τα προβλήματά τους από τις Βρυξέλλες. Και δεν νομίζω πως αυτό είναι σωστό. Και τα δύο είναι λάθος νομίζω. Ε, γιατί ε, κακές εθνικές πολιτικές συνήθως είναι τα που οδηγούν στα προβλήματα και οι λύσεις πρέπει να βρεθούν στο εθνικό επίπεδο. Ε, για να μπορέσουμε λοιπόν να αντιδράσουμε σε, σε, μεγάλα σοκ, όντως θα χρειαστεί ένα εργαλείο σταθεροποίησης όπως έχω πει και παλιότερα, θα μπορούσε να σχεδιαστεί μέσω της χρηματοδότησης ε, το, από χώρε που βρίσκονται σε ε, διαδικασία μεταρρυθμίσεων κτλ. Ε, αλλά ακόμα συζητιόνται, αυτά τα μέσα για το σχεδιασμό, για τον έλεγχο αυτών και είμαστε αρκετά, σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Υπάρχουν πολλές ε, ναι, ε, ενδιαφέρουσες ιδέες. Δεν υπάρχει ακόμα σύγκληση για το θέμα. Ευχαριστώ. Λάγκεν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ανοιχτό και ρεαλιστικό στυλ ε, με το οποίο εργαστήκατε, τώρα παρά τους επένους σας δεν ξέρω εάν ε, ο συναδελφός σας ε, θα μπορέσει να σας διαδεχτεί τόσο εύκολα γιατί είχαμε πάει με την Επιτροπή για τα Panama Papers και ήταν πολύ επιφυλακτικό στην Πορτογαλία κάποια πράγματα τώρα. Είπατε ότι ετέθη το ζήτημα της φορολόγησης της εργασίας. Εμείς ασχοληθήκαμε εδώ πέρα με τη φορολόγηση των κερδών και εκεί πέρα πραγματί τα πράγματα έχουν ως εξής θα ψήσουμε την επόμενη εβδομάδα Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Μάλτα παρά τις εκκλήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται φορολογική παράδοση. Και το πρώτο ερώτημα είναι, το Eurogroup ασχολήθηκε με αυτό το θέμα ή μόνο με τη φορολόγηση της εργασίας. Το δεύτερο ερώτημα είναι άλλο. Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ διαπίστωσε ότι 23% όλων των επιχειρηματικών επενδύσεων παγκοσμίω πρώτα περνάνε από την Ολλανδία. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα άδειών και πνευματική ιδιοκτησίας που έχει μέχρι στιγμής η Ολλανδία είναι ένας λόγος για τον οποίο σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωζώνη έχει κερδισμένους και χαμένους. Συμπτωματικά οι κερδισμένοι είναι όλες οι χώρες εκείνες οι οποίες ε, περιγράφονται ως φορολογικές οάσεις. Αντιθέτως ε, η ε, χαμένη είναι η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος ε, και Ελλάδα. Πώς βλέπετε λοιπόν το μέλλον της Ευρωζώνης, αν συνεχιστεί αυτή η τάση και τι άποψη έχετε για τις ε, τελευταίες προτάσεις της Κομισιόν να μην χρησιμοποιούνται τα κριτήρια του Μαστρίχτη για κάθε χώρα, αλλά συνολικά για την ε, Ευρωζώνη, κάτι το οποίο θα επέτρεπε πιθανώς ε, μεγαλύτερη ανάληψη χρέους κατά 200 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για τη συνεργασία τα τελευταία χρόνια και για και σε εύχομαι καλή επιτυχία για τα, τα φορολογικά. Αυτά από τα γερμανικά μου. Λοιπόν, μιλήσαμε για τα ζητήματα τα φορολογικά, γιατί αν δείτε μακροοικονομικά το ζήτημα, το φορολογικό βάρος στην εργασία είναι πολύ υψηλό. Μόνο η Ιρλανδία έχει πολύ ε, χαμηλή φορολογία της εργασίας, αλλά οι άλλες χώρες είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο του ΩΣΑ και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για το χαμηλότερο μίσο της αγοράς εργασίας. Είναι μια τεράστια πίεση μαζί με την τεχνολογία κτλ. Και ε, βεβαίω ε, υπάρχει μια σύνδεση, δηλαδή αν ήμασταν επιτυχεί στην αποτελεσματική φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων θα μπορούσαμε να μειώσουμε τη φορολογική πίεση στην εργασία. Και συμφωνώ πλήρω με αυτή την προσέγγιση. Κάνατε πολλές ερωτήσεις για την Ολλανδία. Λίγο σε περίεργη θέση γιατί δεν είμαι πια υπουργό Οικονομικών της Ολλανδίας. Α, το ξέρετε, το ξέρετε. Οπότε ε, μπορώ να σας πω το τι κάνει η καινούργια κυβέρνηση, αλλά μάλλον δεν θα έπρεπε γιατί δεν ε, το είναι εκπρόσωπο. Και δεν είμαι σίγουρος ότι και θα μπορούσα να εξηγήσω το τι κάνουν. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Ε, σε γενικές γραμμές ε, προσπάθησα να είμαι όσο δυνατόν ανοιχτός σε αυτό το ζήτημα και αυτό το οποίο κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Τώρα δείχνει η έρευνα του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, κάτι το οποίο ξέρουμε ότι πολλές διεθνείς εταιρείες χρησιμοποιούν το Ολλανδικό φορολογικό σύστημα όχι για να πληρώσουν φόρους στην Ολλανδία, βεβαίως, αλλά για να περάσουν τα κέρδη τους μέσω Ολλανδίας στους πραγματικούς φορολογικούς παραδείσους, ε, στους ε, τροπικούς. Και ελπίζω, θεωρώ ότι αυτό το μοντέλο δεν έχει πλέον μέλλον. Αυτή είναι η απόψη μου. Έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο στην Ολλανδία τα τελευταία πέντε χρόνια, ε, αλλά όχι όσοι θα έπρεπε. Έχουν γίνει πολύ δύσκολες συζητήσεις, είμαι ε, πλέον πολύ ειλικρινής ε, και στον ε, συνασπισμό των δικών μας. Το Εθνικό Κοινοβούλιο στην Ολλανδία δεν είναι υπέρ του να αλλάξει το Ολλανδικό σύστημα, αλλά δεν έχει μέλλον πια. Και αν ε, μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το επιπλέον εισόδημα για να μειωθεί η φορολόγηση της εργασίας, τότε κερδίζουμε και στα δύο μέτωπα. Είναι πολύ πιο δίκαιο. Θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι οικονομίες μας και την ποιότητα ζωής ε, των ανθρώπων. Αυτά. Τι, άλλο να πω. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τους νέους ε, κανόνες ε, για το ευρώ που προτείνει η Κομισιόν ε, την χαλαρότερη μεταχείριση της Ιταλίας και το να παίρνουμε την Ευρωζώνη ως μέσο όρο. Αυτή ήταν πρόταση που δημοσιεύτηκε στο Σπίγκελ. Δυστυχώς δεν ήταν πρόταση της Κομισιόν, λέει ο Πρόεδρος. Ε, το έψαξα στο πακέτο, αλλά... Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας κύριε Πρόεδρε. Διάβασα χτες το πακέτο προτάσεων. Δεν βρήκα κάτι τέτοιο μέσα. Ευχαριστώ, Ιγμπαγέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντάιζελ Μπλουμ, να θίξω και εγώ δύο-τρία σημεία της παρέμβασή σας. Είμαι εισηγητή για την έκθεση την οποία θα πρέπει να ψηφίσουμε σύντομα. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ για τα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε, μολονότι η ανάκαμψη είναι ακόμα αδύναμη. Πάντως οι μακροοικονομικές θετικές εξελίξεις δεν αποτρέπουν τις κοινωνικές ανισότητες σε διάφορες χώρες. Δεν υπάρχει σύγκληση για τα κοινωνικά ζητήματα ανάμεσα στα κράτη-μέλη τη Ευρωζώνης. Αυτό είναι αρκετά αντιφατικό και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της οικονομικής μας πολιτικής. Στο σχέδιο Juncker είχαμε ένα σημαντικό πρωτοβήμα για τον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει όμως να έχουμε και ένα σχέδιο επενδυτικό για τον δημόσιο τομέα. Δεν το λέω εγώ, το λένε πολύ σημαντικοί οικονομολόγοι αλλά και σημαντικοί φορείς στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι θα πρέπει να γίνουν απαραίτητε επενδύσει, Οι υποδομέ μας σε πάρα πολλέ χώρε τη Ευρωζώνης πλέον έχουν παλιώσει. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε το κατάλληλο επενδυτικό κλίμα στον τομέα των μεταφορών, στον ενεργειακό τομέα, προκειμένου να καταφέρουμε να κερδίσουμε και μελλοντικού επενδυτέ. Όσον αφορά δε τι δημόσιε επενδύσει, ακόμα και τι χώρε εκείνε που έχουν δημοσιονομικό χώρο, βλέπουμε ότι οι επενδύσει αυτέ δεν γίνονται. Επομένω, ποια είναι η θέση δική σα και του Eurogroup όσον αφορά το ΑΕΠ τη Γερμανία. Δεύτερη ερώτηση οι ε, φίλοι μας οι Γερμανοί θα έχουν ένα ΕΠ ε, σύντομα δύο φορές ε, υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό θα αποδυναμώσει όμως το ευρώ και κατ' επέκταση και τις εξαγωγές της Ευρωζώνης. Εσείς τι έχετε να προτείνετε σε σχέση με αυτό, σε σχέση με τη δημοσιονομική ικανότητα της Γερμανίας. Και τρίτον, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Λάγκεν για την φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή Μα εξηγήσετε για ποιο λόγο ήταν πολύπλοκο αυτή τη στιγμή να σημειωθεί πρόοδο στο ζήτημα αυτό στα πλαίσια του Eurogroup. Εγώ παρόλα αυτά θα ήθελα να με εξηγήσετε και δυστυχώ τελευταία φορά σα βλέπουμε εδώ πέρα για ποιο λόγο, και δεν το καταλαβαίνω, για ποιο λόγο ορισμένα κράτη-μέλη δεν βρίσκονται σε αυτόν τον μαύρο κατάλογο ή τον γκρίζο κατάλογο όσον αφορά την φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή. Αν δούμε την περίπτωση ε, της Ιρλανδίας και της Apple, η οποία καλείται αυτή τη στιγμή να καταβάλει ένα τεράστιο ποσό, δεν είναι στον κατάλογο αυτό ούτε η δική σας η χώρα, ούτε το Βέλγιο, όπου βλέπουμε εδώ πέρα ότι έγινε μια έρευνα πριν από μερικές μέρες στην πρώην Δέξια, όπου φάνηκε ότι περίπου 3 δισεκατομμύρια είχαν διοχετευθεί σε υπεράκτιες επιχειρήσεις. Αναφέρομαι εδώ πέρα στην Intra Belfius πρώην Για ποιο λόγο δεν βλέπουμε και τη χώρα αυτή στον κατάλογο αυτό. Θα ήθελα για όλα αυτά μια απάντηση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής. Σα ευχαριστώ πολύ. Το να χρησιμοποιούμε μακροοικονομικούς δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης είναι ένας τρόπος να μπορούμε να συνεργαζόμαστε από κοινού διάφορες χώρες και να κινούμεθα από κοινού σε διάφορα διαθροτικά ζητήματα επί των οποίων δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Για παράδειγμα, βιωσιμότητα των συντάξεων. Οι συντάξεις μπορούν να διαφέρουν πολύ από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά σε όλες τις χώρες μας τίθεται το ζήτημα της βιωσιμότητας του εξωτικού συστήματος σε μια κοινωνία ευρωπαϊκή η οποία γυράσκει. Επομένως, οι δείκτες αυτοί συγκριτικής αξιολόγησης έχουν να κάνουν με την εκπόνηση κριτηρίων για την μέτρηση, την αξιολόγηση της βιωσιμότητας, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε πρόθεσμα τη βιωσιμότητα των συντάξεων. Δεν περιγράφουμε ούτε λέμε εμεί εκ των άνω πώς θα πρέπει να σχεδιάζουν τα συνταξιδοτικά του συστήματα τα κράτη-μέλη. Και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον σεβόμενοι την εθνική κυριαρχία για τις πολιτικές εκείνες όπου υπάρχει σαφώς εθνική αρμοδιότητα. Από την άλλη όμως συνεργαζόμενοι μπορούμε να ασκήσουμε ένα στον άλλο πίεση για να κάνουμε τι απαραίτητε βελτιώσει. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, κινούμεθα στα πλαίσια μια νομισματική ένωση. Υπάρχει ο κίνδυνο τη διάδοση προβλημάτων αν δεν θεραπεύσουμε εγκαίρω τα προβλήματα αυτά. Έπειτα, επενδύσει στον δημόσιο τομέα. Αυτό έχει να κάνει με το δημοσιονομικό χώρο. Και ο δημοσιονομικό χώρο δυστυχώ αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζεται στο ίδιο επίπεδο σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωζώνη. Θα ήλπιζα το ζήτημα αυτό να είναι ουσιαστικά πρόσκαιρο Προφανώς η διαφορά αυτή οφείλεται σε μια προβληματική κατάσταση στο παρελθόν. Πιστεύω ότι προϊόντος του χρόνου θα καταφέρουμε να εξορροπήσουμε την κατάσταση και να καταλήξουμε σε ένα ισότιμο επίπεδο δημοσιονομικού χώρου. Αλλά πάλι εγώ θυμάμαι την εποχή που η Γερμανία ήταν ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης και όταν η Γερμανία χρειάστηκε τότε να προχωρήσει σε κάποιες πολύ παρεμβατικές και δύσκολες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας για παράδειγμα. Και βέβαια οι μεταρρυθμίσει αυτέ του κάνουν πάρα πολύ ανταγωνιστικού, του έδωσαν ανταγωνιστικό πλεόνασμα τα τελευταία χρόνια. Θα έλεγα στου Γερμανού φίλου βέβαια ότι α, οι θετικέ αυτέ εξελίξει δεν διαρκούν εσαί. Πρέπει κανεί να είναι πάρα πολύ προσεκτικό με ζητήματα όπω η παραγωγικότητα. Βέβαια θα μπορούσαν άλλε χώρε να αντλήσουν διδάγματα από τη γερμανική εμπειρία ότι είναι σημαντικό να κανεί επαγρύπνηση και να συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομίας της χώρας του. Δεν μπορώ όμω να πάρω τώρα χρήματα εγώ από τον προπολογισμό της Γερμανίας και να τα δώσω αυτά στην Ιταλία και δεν νομίζω ότι τέτοιες μετακινήσεις θα δούμε στο μέλλον. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, και το είπα, είναι αυτή τη στιγμή λύσουμε όλα τα προβληματικά ζητήματα του παρελθόντος μας βαρύνουν ακόμα, να έχουμε τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να αντιμετωπίζουν οι χώρες πιο αποτελεσματικά πιθανούς μελλοντικούς οικονομικούς κλειδονισμούς. Τέλος, όσον αφορά τον ε, μαύρο κατάλογο, πάλι δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το θίξω αυτό. Συζητήθηκε στο ΕΚΟΦΗΝ την Τρίτη. Δεν είμαι όμως πλέον ε, μέλος του ΕΚΟΦΗΝ. Μάλλον θα πρέπει να απευθυνθείτε στον επικεφαλής ε, του ΕΚΟΦΗΝ στα πλαίσια της Εστονικής Προεδρής για να σας πει ποια χώρα έχει ενταχθεί και ποια όχι. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ θετική η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε και όλοι οι συνάδελφοι σας επένεσαν. Ήταν πολύ θετική, επικοδομητική η στάση σας. Εμείς εκτιμούμε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο πάντα υπερασπιζόσασταν τις ιδέες σας, τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο προβάλλατε τις πεπιθήσεις σας. Σήμερα, πέρα από τον εξαιρετικό αυτό τρόπο που εκθέτετε τις ιδέες σας, εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι ήσασταν πάρα πολύ ειλικρινείς Κάνατε μια αποτίμηση του έργου σας, είδατε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Με απόλυτη ειλικρίνεια μας είπατε που είχαμε σημαντικά επιτεύγματα και που ως Ευρώπη σφάλαμε. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν πολύ ειλικρινής και επικοδομητική αυτή η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε και ουσιαστικά συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην δική μας θετική αποτίμηση του έργου σας. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Αγαπητοί συναδελφοί, ας συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Συγγνώμη, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να συνεχίσουμε. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στο 4. Τραπεζική Ένωση, ετήσια έκθεση για το 2017. Ο εισηγητής μας είναι ο Σάντερ Λούνς και θα περάσουμε στην εξέταση των τροπολογιών. 392 τροπολογίες συνολικά κατατέθηκαν. Ο εισηγητής έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλά τα μετρήσατε. Σχεδόν 400 τροπολογίες. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες τροπολογίες τους, γιατί δούλεψαν σκληρά και ε, τώρα είμαστε στη σύνταξη των συμβιβαστικών. Αν δω τις ε, τροπολογίες, βασικά ευθυγραμμίζονται με τις συζητήσεις που είχαμε εδώ στις 9 Νοεμβρίου. Κάποια γενικά σχόλια για τις τροπολογίες. Σημείωσα ότι πολλές ε, είναι συνυπογεγραμμένες από την κυρία Χούμπνερ και την κυρία Ντελβό για όσους πιστεύουν ότι έχει πεθάνει ο Μέγας συνασπισμός μετά την άφηξη του κυρίου Ταγιάννη, ε, ξυπνήστε. Πιο σοβαρά όμως αυτές οι συνυπογεγραμμένες τροπολογίες μας δίνουν την αίσθηση της ατμόσφαιρας που επικρατεί στην αίθουσα και θα μας διευκολύνει να βρούμε ευρείες συνενετικές λύσεις για κάποιες ε, υποθέσεις, αλλά ήταν αστείο που το, το διαπιστώσαμε. Τώρα έχουμε μια όχι και τόσο πολιτική γραμμή. Άλλες τροπολογίες νομίζω αντικατοπτρίζουν περισσότερο τις γραμμές του ίδιου του τραπεζικού τομέα. Έχουμε λοιπόν διάφορες ιδέες. Πάντοτε καλό είναι να είμαστε σύντομοι και περίκτικοι. Ίσως λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την έκθεση, αν και η εμπειρία μας δείχνει ότι αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο. Ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να μιλήσω για τις δικές μου τροπολογίες γιατί στις 9 Νοεμβρίου εγώ ε, επέλεξα να παρουσιάσω μια ουδέτερη έκθεση και μετά επέβαλα και κάποιες τροπολογίες για κάποια σημεία που θα ήθελα να προσθεθούν. <coughs> να αναφέρω ότι οι κίνδυνοι των εθνικών τραπεζικών συστημάτων δεν αντιμετωπίζονται αρκούντος και ανέφερθηκα στην ε, Banca στη Βένετα, στην, ε, στο Banco Popular και διάφορες άλλες τράπεζες, τη Βιτσέντς και τα ε, επίσης έχω το, το αντέντομ της ΕΚΤ στις κατευθυντήριες της γραμμές, είναι λεπτό το θέμα. Ξέρω ποια είναι η γνώμη της νομικής υπηρεσίας και θέλω να τονίσω εδώ στην Επιτροπή ότι επίσης ε, συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εκφράζονται σε εκείνη την έκθεση. Γνωμοδότηση μάλλον. Ακόμα Πρέπει αναφέρομαι στον κίνδυνο όσον αφορά τη συγκέντρωση κυρίω ομολόγων γιατί συσχετίζεται με το κρατικό χρέο αυτό και για άλλα θέματα αναφέραμε στο κεφάλαιο και την ρευστότητα άρθρα 6 και 8 της CCRR. Έχα και κάποιες παρατηρήσεις για τις σχετικές ενισχύσεις και τα λοιπά. Όλες αυτές οι ιδέες βεβαίως θα συζητηθούν ανοιχτά στις συνεδριάσεις των σκιωδών, πρώτη εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Τρίτη στο Στρασβούργο. Και ε, Βέβαια έχουμε και κάποιες τρομεπολογίες που πιστεύω πως πρέπει να σεβαστούμε την εργασία της κυρίας Δελάγκε και ε, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και την εργασία μας σε αυτές τις συνεδριάσεις. Τώρα για το χρονισμό δουλεύουμε σκληρά για να συντάξουμε τις συμβαστικές, θα σας τις στείλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και η πρώτη ε, συνεδρία των σκιωδών είναι την τρίτη όπως σας είπα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Εκτιμώ. Το γεγονό ότι είστε πιεσμένοι χρονικά το γνωρίζουμε και από πέρι, τα προηγούμενα χρόνια ότι έτσι το χρον, η προθεσμία είναι ενδεικτική. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι ντε και καλά να το υποβάλουμε στις 24 ε, Ιανουαρίου. Αυτό για να σας ανακουφίσω κάπως. Και τώρα. Τώρα για τις συμβιβαστικέ να είναι πολλές και σας ευχαριστώ που κάνετε τον κόπο να τις επιτύξετε σε συμβιβαστικέ. Πολύ καλή η επικοδομητική αυτή προσέγγιση. Και τώρα περνάμε στους κοιόδης. Ε, ξεκινάμε με τον Εξ ονόματος των ε, συνυπογραφών να πω η Δούντα δεν μπορούσε να είναι εδώ, ε, μου ζήτησε να πάρω εγώ το λόγο εξ ονόματός της και προσβλέπει στη συνεργασία μαζί σου. Τα βασικά σημεία είναι ότι έχουμε δύο κύριες αρχές. Στι τροπολογίε. Το πρώτο είναι να αποφύγουμε οποιαδήποτε σύσταση ιδιαίτερα περιγραφική που να αφορά τις, ε, τους φακέλους που, δεν, που, είναι υποδιαπραγμάτευση. Αυτή την προσέγγιση ακολουθήσαμε πέρυσι και Θέλουμε να την συνεχίσουμε. Δύο χρόνια συζητάμε αυτό το θέμα. Η Κομισιόν θέλει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Το τραπεζικό πακέτο θα αρχίσει να συζητιέται την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε σε κρίσιμη φάση για τους νομοθετικούς φακέλους. Δεν θέλουμε να προκαταβάλουμε ε, την εργασία που γίνεται αλλού. Τώρα, παράγραφοι 22, 21 και παράγραφες, παράγραφη 6 ε, στις ε, εκθέσεις που φορούν την, ε, C, την ERC, e την ε, ERCD και τα λοιπά. Δεύτερη κατευθύνη γραμμή είναι να αποφύγουμε να καταδείχνουμε συγκεκριμένους θεσμούς. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας, το έχουμε συμφωνήσει στην έκθεση πέρυσι. Είπαμε ότι θα λαμβάνουμε υπόψη τις εκθέσεις των ε, ειδικών επιτροπών όπως οι δύο διαδοχικές τάξεις. Αποφύγουμε λοιπόν την αναφορά συγκεκριμένων θεσμών. Τώρα για τα σχόλια επιμένουμε για τις όρους ε, όπου υπάρχουν ε, Κοινές ε, εποπτικές ε, λειτουργίες από πλευράς ΕΚΤ και εποπτικών αρχών και με τον ε, SRB και για τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, Εποπτικής Αρχής και των κρατικών εποπτικών αρχών, οι εποπτικές αυτές αποφάσεις είναι, μπορούν να λαμβάνονται κοινά. Επίσης ζητούμε να υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση για τα θέματα του ε, και των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά ο κίνδυνος για δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και η ΕΚΤ έχουν αρχίσει να εργάζονται για αυτό το θέμα και γι' αυτό είναι σωστό να πούμε ότι χρειάζονται περαιτέρω ενέργεια σε όλα τα επίπεδα. Επίσης θυμίζουμε την ανάγκη να φροντίσουμε να μην αυξηθούν τα κεφάλαια γενικώ ε, υπό το φως της ολοκλήρωσης Βασιλείας 3 αλλά και υπό το φως των όσων θα ε, εκδοθούν κρατικά ομόλογα ή όχι και ε, επίσης κατά πόσο με τα, με τα χρεόγραφα θα οδηγηθούμε σε αμοιβιοποίηση και τα λοιπά. έχουμε και στοιχεία για τις συγκεκριμένες επιπτώσεις ε, στον ε, τραπεζικό τομέα και οι τράπεζες θα πρέπει να είναι έτοιμες να ε, δεχτούν τις αλλαγές που προβλέπονται. Έχουμε και τις κανόνες αφαιρεγγιότητας που εφαρμόζονται και για τις τράπεζες. Οι τράπεζες αυτές είναι ένας μεγάλος πληθυσμός, μεγάλο κομμάτι του τραπεζικού πληθυσμού και αν δεν εναρμονιστεί αυτή η πτυχή δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ισότιμο πεδίο για τις τράπεζες σε ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση. Αγγίζουμε τα προβλήματα που που προκαλούνται από τις διάφορες κρατικές ε, επιδοτήσεις λόγω της εξυγίανσης ε, ε, άλλων λειτουργιών. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση. Επίσης θυμίζουμε ένα θέμα όπου ο πρόεδρο τη Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων η Ντανούτα το έχει ε, δουλέψει και μάλιστα έχει γίνει και σχετική ε, συζήτηση για το πώς το Fiscal Pact θα μπει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έπειτα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έντονη γλώσσα στο για τον προστατευτικό ε, μηχανισμό θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σχετική εργασία μόλις αυτό είναι εφικτό. Εξ ονόματος λοιπόν της ε, Ντανούτα που δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι σήμερα παρούσα, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας στη διάρκεια των ε, συνεδριάσεων των σκιωδών που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα και ελπίζουμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα και σας ευχαριστώ πολύ. Τι έχει να κάνει το Fiscal Compact με την ε, Τραπεζική Ένωση. Δεν κατάλαβα ακριβώ. να ξαναδιαβάσω την τροπολογία, μπα και καταλάβω. Λέει ο πρόεδρο. τελεβό, ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να αναφέρω ότι προφανώς οι τροπολογίες που έχουμε συνυπογράψει οι υποφαινόμενοι και η Ντανούτα Χούμπνερ είχαν ως στόχο να διευκολύνουν τον εισηγητή διότι βασίσαμε την ε, μεταξύ μόν συνεργασία στις δύσκολες, πολύ δύσκολες συζητήσεις που κάναμε πέρυσι για την περσινή ετήσια έκθεση για Τραπεζική Ένωση και είδαμε ότι υπήρχαν σημεία επί των οποίων επί της αρχής είχαμε συμφωνήσει πέρυσι και είπαμε ότι για τα σημεία αυτά θα μπορούσαμε ήδη από τώρα να έχουμε μια κοινή στάση. Σε καμία περίπτωση θέλαμε βέβαια εμεί να προδικάσουμε τη γενικότερη μορφή της έκθεσης, γιατί θα έπρεπε να εκφραστούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένε αναφορέ στην έκθεση στα ζητήματα αυτά επί την οποία υπάρχει συμφωνία. Επίση, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να ισχύει αυτό το οποίο είπαμε και πέρυσι. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει αν λοιπόν πέρυσι σε κάποια σημεία είχαμε μια πιο πολύπλοκη διατύπωση και αν καταφέραμε τελικά να καταλήξουμε πέρυσι κάποιο συμβασμό, ε, θέλαμε να ενσωματώσουμε το συμβασμό αυτό και στη φετινή έκθεση. Όσον αφορά τώρα το αν μπορούμε να κατονομάσουμε συγκεκριμένες χώρες, εταιρείε, οντότες κτλ. Λέμε εμεί ότι θα πρέπει περισσότερο να δούμε τα πράγματα πιο σφαιρικά και γενικά, να δούμε που υπάρχουν αποτυχίες και αδυναμίες, που βάλουν κατά του γενικού συμφέροντος, χωρίς όμως να υπάρχει λόγος να κατονομάζουμε συγκεκριμένες τράπεζες. Και γι' αυτό σε όλους τους λόγους λοιπόν συνυπογράψαμε τις τροπολογίες αυτές. Βλέπουμε όμως ότι οι συνάδελφοι δεν συμφωνούν αναγκαστικά με όλες αυτές τις τροπολογίες. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες άλλες τροπολογίες, οι οποίες, ενδεχομένως, να είναι και κάποιες προβληματικέ, γιατί όπως είπα και την προηγούμενη φορά, Το προήμιο της έκθεσης ήταν ιδιαίτερα απεσιόδοξο. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν αν μη τι άλλο κάποια αισιόδοξα στοιχεία γιατί μία κάποια πρόοδο την έχουμε σημειώσει στην Τραπεζική Ένωση. Όσον αφορά την εποπτεία, θεωρώ ότι θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο γιατί μόνο μέσω της εποπτείας μπορούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε κάποιο λόγο. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε κάποια πιο πρακτικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διασφαλίσουν οι χώρες προκειμένου και εμείς να μπορούμε να έχουμε κάποιο λόγο. Εμένουμε μέσω τροπολογιών περισσότερο στο FinTech, όλη αυτή την νέα τεχνολογία των τραπεζών. Επίσης, τα προληπτικά τα προληπτικά, μακροπροληπτικά με συγχωρείτε εργαλεία δεν επαρκούν και όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εμένουμε εδώ πέρα στην ευθύνη που φέρουν τα κράτη-μέλη, αλλά λέμε παράλληλα ότι θα πρέπει δράση να ληφθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ χρησιμοποίησα τη συγκεκριμένη μάλιστα τροπολογία για να κάνω και ένα γενικό σχόλιο για το ευνομοθετήν, για την καλύτερη δυνατή δηλαδή νομοθεσία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε δηλαδή τις αρχές της διαφάνειας, θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση, αξιολόγηση αντικτύπου και για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά και για την νομοθεσία στο τρίτο επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά θα στείλει το σωστό μήνυμα προς, τους, προς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Τούτων λεχθέντων μπορούμε να δείξουμε ένα επικοδομητικό πνεύμα και νομίζω θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. ότι η Κονιγέ δεν είναι στην αίθουσα. Κανείς από τους φελεύθερους μάλιστα. Βιέγκας παρακαλώ. Καλημέρα σας. Θα μιλήσω πορτογαλικά όπως συνηθίζω. Το να μιλάμε για αυτή την ετήσια έκθεση για την Τραπεζική Ένωση σημαίνει ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν, ποιοι ήταν οι στόχοι που διέπουν την ιδέα της δημιουργίας της Τραπεζικής Ένωσης. Να αποφύγουμε τη χρήση δημόσιου χρήματος για την διάσωση των τραπεζών, αλλά και να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο των πολύ μεγάλων τραπεζών για να πτωχεύσουν. Αλλά από αυτό το πρίσμα να το δούμε νομίζω πως κάνουμε το αντίθετο στην Πορτογαλία και όχι μόνο ε, όπου παρακολουθούμε τη συνεχή χρήση δημόσιου χρήματος για την προστασία των χρεών ε, για την χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και από την άλλη πλευρά παρακολουθούμε επίσης φαινόμενα συγκέντρωσης που οδηγούν στο να υπάρχουν και μέχρι σήμερα, ε, υπάρχει μάλλον σήμερα ένας ε, χρηματοπιστωτικός τομέας εξαιρετικά συγκεντρωμένος και αυτό προκαλεί ε, θεμητές αμφιβολίες. Δηλαδή, αν έχουμε το πολιτικό σθένος για να επιβάλλουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες γιατί είναι προφανές ότι το χρηματοπιστωτικό λόμπι μαζί με τα κρατημέλη, μαζί με τις κυβερνήσεις, μαζί και με τα κόμματα που υπερασπίζονται τα συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού τομέα ε, αντιστέκεται και κάνουν λιγμούς για να ελαχιστοποιήσουν ακόμα και να κυρώσουν ή να εξουδετερώσουν το σύνολο των νομοθετικών μέτρων που από άποψη ε, ε, οικονομική έχουν νόημα. Στην πράξη βέβαια η εφαρμογή τους δεν αντιστοιχεί σε αυτό που θα αναμέναμε. Πιστεύω πως το θέμα της διάλυσης της, της μάλλον της ε, Banco Popular είναι αναπαυκτό και είχε φέρει στο φως όλες τις αδυναμίες του τομέα, την ελληπή εποπτεία, στην, ε, πώς το έχει χειριστεί και η Ιταλική Κεντρική Τράπεζα, αλλά δείχνει και τις, τα δικά μας λάθη, γιατί μάθαμε ότι το σύστημα εξωτερικεύει στην πράξη την εποπτεία. μαζί με τους μεγάλους ε, τέσσερις, τις μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες που τα τελευταίες δεκαετία ε, εξοραίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εκεί προστρέχει η Τραπεζική Ένωση ώστε να κάνει την υποπτία και να βασίσει σε, αυτές, σε αυτά τα στοιχεία της αποφάσης της για την τραπεζική εξηγήση και αυτό τελικά οδηγεί σε μια αρνητική εκτίμηση τη ε, Τραπεζική Ένωση το τελευταίο χρόνο και ενισχύει την βασική μα θέση για αυτό το θέμα, ότι δηλαδή τελικά θα έπρεπε να στοχεύσουμε στην πιο εύκολη λύση και την πιο προφανή, ότι θα πρέπει δηλαδή να βασιστούμε στο δημόσιο χρηματοπιστωτικό τομέα που είναι πραγματικά στην υπηρεσία των ανθρώπων και τη οικονομία. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω εδώ τους πράσινους οπότε EFDD Μάρκο Βάλλη όχι Αρμπαράκα Any catch request Θέλει κάποιος τον λόγο στο catch the eye Παρακαλώ λοιπόν ο εισηγητής Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ε, σκιώδης εισηγητές και αναμένω και τις ε, συναντήσεις μας, πρώτη συνάντηση την Τρίτη. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε τις τροπολογίες των συντομότερο δυνατών. Κάποια πράγματα για τον... το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευελιξία σας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα καταφέρουμε εντός του χρόνου και είμαι σίγουρος ότι με το προσωπικό μας και τους ε, συμβούλους ε, του ECR ε, θα τα καταφέρουμε. Τώρα, για την σχέση με την Τραπεζική Ένωση έχω και εγώ την ίδια παρατήρηση με εσάς, αλλά εάν αφήσω ελευθερή την δημιουργικότητα δεν ξέρω αν θα έρθουμε πιο κοντά σε συμβασμό. Τώρα για τις σοσιαλδημοκράτες και το ότι δεν θέλουν να, να κατονομάσουμε άτομα ε, είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν το ακολουθήσουμε σε όλες τις εκθέσεις ε, της Επιτροπής μας θα είναι οπωσδήποτε ενδιαφέρον ε, γιατί έχουμε και το θέμα του ανταγωνισμού, αλλά τέλος πάντων περιμένω τις συζητήσεις αυτές. Επίσης, για την κυβερνοασφάλεια. Αυτή είναι πολύ καλή πρόταση των σοσιαλδημοκρατών και αναζητούμε συμβαστικές ε, τροπολογίες και εκεί για να προσθέσουμε κάτι και το να προσθεθούν νέες ιδέες στην έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε... Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. Όπως ξέρουμε, είναι ενδεικτικά όλα 24 Ιανουαρίου, στην περίπτωση στην Ολομέλεια αλλά θα ακολουθήσουμε την αξιολόγηση της διαπραγματευτικής ομάδας. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Υποχρεωτική... Ναι, υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σε σχέση με διασυνορικές ρυθμίσεις. Ε, ο εισηγητής είναι ο Εμμανουέλ Μόρελ. Έχετε τον λόγο. Euh, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι τα φορολογικά σκάνδαλα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι Ευρωπαίοι πολίτες εντελώς θεμητά πλέον και δικαιολογημένα θεωρούν ότι υπάρχει μια πλήρης ατιμορρησία για πάρα πολλές επιχειρήσεις, για εταιρείες holding, για πολυεθνικές, οι οποίες καταφέρνουν μέσω μηχανισμών που βρίσκονται στα όρια του νόμου να παρακάμπτουν τους, τις φορολογικές αρχές και τελικά να μην καταβάλουν φόρους. Το ζήτημα αυτό βέβαια πάντα ξεπερνούσε το εφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο γιατί όλες οι εκθέσεις που εγκρίναμε στο παρελθόν ζητούσαν απόλυτη διαφάνεια, διαφάνεια στις εμπορικές συμφωνίες που συμνάπτουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και Έπειτα είχαμε την οδηγία αυτή, την οποία σας παρουσιάζουμε σήμερα, που αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές τελικά πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διορθωθούν τα κακό κείμενα. Γιατί ουσιαστικά ασχολούμεθα εδώ πέρα πιο συγκεκριμένα με τους ενδιάμεσους και συγκεκριμένα με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Υπάρχει μία πραγματική βιομηχανία, ένας πραγματικός κλάδος επαγγελματικός αν θέλετε, για την παράκαμψη των φρολογικών κανόνων. Δικηγορικά γραφεία, γραφεία παροχής συμβουλών, πάρα πολλοί άνθρωποι ουσιαστικά που έχουν ως στόχο να συμβουλεύσουν συγκεκριμένε επιχειρήσει επιχειρήσεις για τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να παρακάμψουν τις φορολογικές υποχρεώσεις. Το είδαμε αυτό και στο πλαίσιο των Paradise Papers και στο πλαίσιο των Panama Papers. Έχουμε πλέον ένα κατάλογο πολύ μεγάλο και διεξοδικό για τους μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορισμένες επιχειρήσεις προκειμένου να παρακάπτουν τη φορολογία. Στα πλαίσια λοιπόν της νέας προτινόμενης οδηγίας καλούμεθα κάθε φορά να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάθε μία τέτοια νέα μέθοδο η οποία επινοείται και χρησιμοποιείται για την αποφυγή των φορολογικών υποχρεώσεων. Σε όλα αυτά λοιπόν αναφέρεται η προτινόμενη αυτή οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία θεωρώ ότι μπορούμε να χαιρετήσουμε. Θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε και κάποιες βελτιώσεις. Ήδη εγώ έχω κάποιες πρώτες ιδέες, οποίες θα μπορούσα να συζητήσω με τους σκιώδεις ηγητές. Βελτιώσεις που ουσιαστικά ανταποκρίνονται και στις δικές μας προσδοκίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο φορολογικό τομέα. Η πρώτη βασική αλλαγή η οποία προτείνω είναι ίσονο ενδεχομένω σημασία, αλλά σημαντική από την άλλη είναι σημαντικό για παράδειγμα να γίνεται μία αναφορά στους πραγματικούς δικαιούχους των καταπιστευματικών ταμείων. Δεν γίνεται τέτοια αναφορά αυτή τη στιγμή στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε κυρώσει για όλους αυτούς τους ενδιάμεσους, οι οποίοι δεν εμφανίζονται στις εκθέσεις που βάλουν τα κράτη-μέλη και όχι μόνο θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, αλλά κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι χρηματικές. Δεν μπορούμε ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε ευνοϊκά τους ανθρώπους αυτούς όταν παραβαίνουν τους κανόνες. Και λέμε επίσης ότι σε σχέση με την πολιτική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος έλεγχος για τα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο έλεγχος αυτός βέβαια θα καταστεί δυνατός μόνο αν τα κράτη-μέλη παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια απόλυτης εμπιστευτικότητας όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διεξάγει τους απαραίτητους ελέγχους να γίνονται διαθέσιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς στιγμή, η υφιστάμενη οδηγία καλύπτει ε, τους μελλοντικούς κανόνες, μελλοντικούς αν θέλετε διασυνοριακούς διακανονισμούς αποφυγής ε, καταβολή των φόρων, νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά κρίμα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, πολλές επιχειρήσεις ή καταπιστευματικά ταμεία τα οποία χρησιμοποιούν ε, τεχνάσματα φορολογικά τα οποία επινοήθηκαν για παράδειγμα πριν από ένα χρόνο, πριν από πέντε-δέκα χρόνια και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις φορολογικές αρχές να γνωρίζουν ότι υφίστανται αυτές οι οντότητες γιατί ε, όσο πιο πολύπλοκα είναι τα τεχνάσματα αυτά τόσο μεγαλύτερη είναι και η απάτη που επιτελείται πίσω από τα τεχνάσματα αυτά. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να καλύψουμε όχι μόνο τις μελλοντικές αυτές διασυνοριακές ρυθμίσεις, αλλά και τις ήδη υπάρχουσες, τις παρελθούσες. Να δούμε δηλαδή ποιο είναι, αν θέλετε, το απόθεμα, το σωρευτικό τέτοιων φορολογικών τεχνασμάτων και ρυθμίσεων που έχουμε ήδη μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να καταγγελθούν και αυτές οι ήδη φυστάμενες περιπτώσεις. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, η κοινή γνώμη, έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες από εμά στο ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να σταματήσουμε να διεξάγουμε ένα φορολογικό πόλεμο μεταξύ κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, θα πρέπει να καταφέρουμε να ανοιχνεύσουμε και να εντοπίσουμε όλα αυτά τα κέρδη τα οποία φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να φορολογούνται. Θα πρέπει επίση να καταρρύψουμε όλα αυτά τα τεχνάσματα φορολογική βελτιστοποίηση και αποφυγή καταβολή των φόρων. Και τέλο, να καταφέρουμε τελικά να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα καταβολή των φόρων προ το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό θα πρέπει να γίνει μια πραγματικότητα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει βέβαια ακόμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Φλούβιο Μαρτουτσέλο έχει το λόγο, εξ ονόματος του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στόχος μας εδώ πέρα είναι να καταφέρουμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες του φορολογικού ελέγχου και να αποφύγουμε φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και να καταφέρουμε να έχουμε περισσότερες και πιο ποιοτικέ πληροφορίες που αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή. Θα μπορούσα να συμφωνήσω με αρκετά σημεία, θα πρέπει αυτά να τα επεξεργαστούμε περισσότερο να δούμε στις συζητήσεις των σχεδόν εισηγητών πώς τα βελτιώσουμε. Υπάρχουν άλλα σημεία με την οποία δεν συμφωνούμε. Το, η τροπολογία 1, όπως και η τροπολογία 20, είναι τροπολογίες με τις οποίες δεν μπορεί να συμφωνήσει το ΕΛΚΑ, γιατί αναφερόμαστε εδώ πέρα σε μια φορολογική ισότητα, φορολογική δικαιοσύνη και ότι θα έπρεπε ουσιαστικά αυτό να επιτευχθεί μόλον ότι υπάρχουν διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές και όσον αφορά την τροπολογία 3. Πρέπει εδώ πέρα η αρχή που προβλέπεται να αντιστραφεί. Έπειτα, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή το οποίο έχουμε στην τροπολογία 7, πρέπει να εξετάσουμε λίγο εδώ πέρα περισσότερο τις λεπτομέρειες στην συνεδρίαση των συντονιστών. Ακόμα και η πρόταση αναδρομικής ισχύς για 14 χρόνια νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε λίγο περισσότερο. Αυτό προβλέπεται στην τροπολογία 10. Για την τροπολογία 12 προτιμούμε το αρχικό κείμενο όσον, όσον αφορά την διάχυση των εμπορικά απόρριτων πληροφοριών. Πολλές προτάσεις επιθυμούμε να κάνουμε προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα ελέγχου και προσβλέπουμε σε μια θετική συνεργασία προκειμένου να έχουμε έναν μηχανισμό ακόμα πιο αποτελεσματικό. Σας ευχαριστούμε. Πύρκο Ροκόνεν Λέρνερ από το Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ε, προηγούμενους ομιλητές. Ε, η πρόταση αυτή είναι πολύ φιλόδοξη. Τα παραθυράκια τα βρίσκουν ε, αυτοί γρηγορότερα από όσο οι νομοθέτες τα κλείνουν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η πρόταση αυτή επιτρέπει και υποχρεώνει λογιστές, δικηγόρους, τραπεζίτες να ειδοποιούν αμέσως στις αρχές όταν παρακολουθούν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και επειδή οι πληροφορίες βεβαίως ε, θα κυκλοφορούν μεταξύ των κρατών μελών αυτό σημαίνει πως οι φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών να διορθώσουν την κατάσταση ακόμα και εντός του τρέχοντος ε, φορολογικού έτους. Ακόμα λοιπόν και αν, ε, αν είχε εφαρμοστεί αυτή η κατάσταση θα είχε αποφευθεί η κατάσταση στην Ιρλανδία με την Apple. Η Κομισιόν θεωρεί ότι τα προληπτικά μέτρα επαρκούν γιατί οι εταιρείε φοβούνται για τη φήμη τους. Όμως, αν δεν δημοσιευτούν αυτές οι πληροφορίες αλλά τις μοιραστούν μόνο οι φορολογικές αρχές, δεν θα πληγεί η φήμη των εταιριών. Επίσης, θα πρέπει να ερευνηθούν οι εταιρείε για να προληφθεί η φοροδιαφύγη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι χώρες οι οποίες προσελκύουν εταιρείε με χαμηλά επίπεδα φορολογίας όπως η Ιρλανδία ε, θα πρέπει να έχουν επαρκή συστήματα για να, να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή. Είναι πολύ σημαντικό όλες οι χώρες να έχουν επαρκή συστήματα για να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα μπορούν εύκολα να παρακολουθούν οι φορολογικές αρχές και να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση. Είναι σημαντικό να μπλοκάρουμε όλα τα πιθανά παραθυράκια έτσι ώστε οι μεγάλες εταιρείες όπως η Apple να πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί εγκαίρως. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Λιβ Βιέρνιχ. για την Κύριε Μορέλ, σας ευχαριστώ για την δουλειά που κάνατε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την στήριξή μου για την πρόταση της Κομισιόν. Πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί ένα πεδίο ισοανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών και να υπάρχει και διαφάνεια για να διασφαλίσουμε τα φορολογικά μας έσοδα τα επόμενα έτη. Όμως, όπως επισημαίνει ο εισηγητής, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν και κάποια που πρέπει να διευκρινιστούν. Κυρίως η απόφαση της ε, Κομισιόν να ασχοληθεί μόνο με μελλοντικέ τέτοιες διευθυντήσεις. Βεβαίως υπάρχει αρχή της μία αναδρομικότητας που πρέπει να γίνει σεβαστή. Πρέπει να αποφύγουμε την νομική αβεβαιότητα. Όμως, όπως επεσήμανε ο εισηγητής, συστήματα τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή δεν θα εμπιθούν στην νέα οδηγία και άρα θα υπάρχει καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων. Έχοντας κατά νου ότι το διοικητικό βάρος ε, στους ενδιάμεσους πρέπει να παραμείνει στο ελάχιστο, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί την προσοχή μας ε, και έτσι πρέπει να ε, το συζητήσουμε περαιτέρω. Επιπλέον, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ασφάλεια των ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών. Τέλος, άκουσα ότι κάποιοι θεωρούν ότι ε, το όλο αυτό σύστημα και η διάταξη είναι πολύ ε, γενικόλογη και όχι αρκετά συγκεκριμένη και οδηγεί σε νομική ανασφαλεία. Από την μία αντιλαμβάνομαι αυτές τις ανησυχίες, από την άλλη δεν, επιτρέ... δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε νέα παραθυράκια με το να γίνουμε πολύ συγκεκριμένοι, αν έχουμε προτάσεις οι οποίες συμμορφώνονται και με τις δύο αυτές απαιτήσεις. ευχαριστώ να τις συζητήσω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ ο κύριος Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον συνάδελφο Εμμανουέλ Μορέλ, για την ε, δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα και να πω ότι δεν μπορούμε να συζητούμε αυτή την πρόταση με το πνεύμα business as usual, γιατί είμαστε στο φως των αποκαλύψεων των Paradise Papers που έχουν ανεβάσει στην κορυφή της ατζέντα αυτήν την εγκληματική και μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή. Και το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Πώς μπορούν μερικές εκατοντάδες δημοσιογράφοι να βρίσκουν περισσότερα στοιχεία εναντίον αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας από ότι τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο, η Κομισιόν, οι διεθνείς μηχανισμοί. Η Κομισιόν λέει ότι είναι στις προτεραιότητες της ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Αλλά τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι πενιχρά. Η Διεύθυνση Ερευνών και Μελέτης του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτιμάει με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς ότι κάθε χρόνο χάνουν τα κράτη-μέλη και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός από 50 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και αυτό σημαίνει υπερφορολόγηση των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επειδή κάποιες πολυεθνικές με τη βοήθεια τραπεζών και ειδικευμένων ε, δικηγορικών εταιριών παραβιάζουν τους κανόνες της χρηστής διαχείρισης και της δίκαιης φορολογίας. Εγώ σε αντίθεση με τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ορισμένες συμπαθείς γενικότητες που άκουσα από την εισηγήτρια των φιλελευθέρων, θα ήθελα από τον εισηγητή τον κύριο Μορέλ να κάνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένες προτάσεις για να περιορίσουμε τα περιθώρια των πολυεθνικών να εγκληματούν εις βάρος του κοινωνικού κράτους, των κρατικών προϋπολογισμών και όλων των υπολείπων φορολογουμένων, οι οποίοι είναι το 99,99% των κοινωνιών μας και των ψηφοφόρων μας, τα πρόσθετα όλων των πολιτικών ομάδων και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Φιλελευθέρων. Και εδώ χρειαζόμαστε φορολογική εναρμόνιση, υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών, αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες και όλοι ξέρουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτό το θέμα, αυτή η μέγα φοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνική κλίμακα. Τα, τα περιθώρια σε εθνική κλίμακα είναι περιορισμένα. Χρειάζεται ευρωπαϊκή συνεργασία, ισχυροί κανόνες και να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο G20 να θέσει αυτά τα θέματα. Και όταν συζητάμε για φορολογικούς παραδείσους, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φορολογική παράδειση δεν υπάρχουν μόνο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι το ξέρουμε αυτό. Επομένως είμαι ε, διατεθειμένος να συνεργαστώ με τον εισηγητή και θα ήθελα αυτά που λέμε γενικά, ότι είναι κακό πράγμα η φοροδιαφυγή και είναι σκανδαλώδες αυτό που αποκαλύπτουν τα Paradise Papers, όταν έρχονται συγκεκριμένες προτάσεις για τον περιορισμό, να το υποστηρίζουμε με συνέπεια. Αλλιώς θα διαιωνίζεται η φοροδιαφυγή με, τις δικές μας, με τη δική μας ανοχή και συνευθύνη. Thank you. Σας ευχαριστώ. Σκοτ Κέιτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συγχαρώ και εγώ με την σειρά μου τον κύριο Μορέλ και στηρίζουμε σε γενικές γραμμές ε, το σχέδιο που έχει υποβάλει. Η Κομισιόν έκανε μια πρόταση για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και θεωρούμε ότι πρέπει να εγκριθεί το μόνο δυνατόν. Επίσης συμπίπτει με το σχέδιο BEPS, ε, το σχέδιο δράσης του ΟΣΑ, οπότε θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ηγηθεί στην διεθνή μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Υποστηρίζουμε την πρόταση του εισηγητή να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής ε, των συμφωνιών που πρέπει να αποκαλυφθούν, ε, τα σημεία 5 και 6 και των ενδιάμεσων ε, που δεν είναι μόνο τα άτομα τα οποία είναι φορολογικοί σύμβουλοι, αλλά οποιοδήποτε δεν είναι τέτοιες συμβουλές και επίσης χρηματοοικονομική συμβουλή κτλ. Επίσης θα πρέπει να καταρτιστούν κατάλογοι για τα συστήματα τα οποία απαγορεύονται από τα κράτη-μέλη, γιατί αυτά θα χρησιμεύσουν στους επαγγελματίες για να ξέρουν το τι απαγορεύεται και τι όχι. Τώρα για το σημείο 10 δεν ξέρουμε γιατί υποστηρίζει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα συστήματα από το 1993. Εμείς θα υποβάλουμε μια σειρά τροπολογιών, πρώτα μια σύσταση προς τα κράτη-μέλη για να επεκτείνουν την υποχρέωση αποκάλυψης και για συστήματα που λειτουργούν και σε μία μόνο χώρα. Αυτό υπάρχει ήδη και, μια, και ως σύσταση της Επιτροπής ε, Πάναμα. Επίσης, μιλάμε εδώ πέρα για διασυνοριακές καταστάσεις, δηλαδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος η Κομισιόν δεν έχει νομική βάση να υποχρεώσει ενδιάμεσους να αποκαλύψουν συμφωνίες που ισχύουν μόνο σε χώριο επίπεδο αλλά θα πρέπει να το καλύψει το μέλλον. Για την αναδρομική δημοσίευση συμφωνιών, η τρέχουσα συμφωνία λέει ότι η αποκάλυψη φορολογικές αρχές θα ξεκινήσει μόνο όταν έχει γίνει η Διεθνές δίκαιο Οδηγία του 2019, αλλά οι ενδιάμεσοι θα πρέπει να αποκαλύψουν ε, αναδρομικά από την δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε συμφωνία ε, εμείς ε, καλύπτεται από την πρόταση και είναι ακόμα ενισχύ θα πρέπει να αποκαλύπτεται χωρίς ε, χρονικό όριο αλλά επίσης θα μπορούσαμε να δούμε το χρονικό όριο των 5 ετών με τον εισηγητή για τις ανταλλαγές πληροφοριών θεωρούμε ότι στο μέλλον τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να υποβάλλονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων που θα είναι προσβάσιμη από όλα τα κράτη-μέλη. Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να τεθεί ενισχύ νωρίτερα από όσο προτείνει η Κομισιόν. Το κείμενο λέει μόνο θα μπορούσε ή θα έπρεπε. Εμεί θέλουμε δεσμευτική υποχρέωση. Η πρόταση θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξη αν περιείχε μια υποχρέωση για τους ε, όρκωτους έλεγκτες ε, ε, να αποκαλύπτουν τέτοιες περιπτώσεις όταν υποπίπτουν στην αντίληψή τους και τέλος θα επανέλθουμε στο γνωστό που λέμε πάντα ότι πρέπει να επενδύσουν περισσότερα τα κράτη-μέλη στις φορολογικές τους διοικήσεις γιατί θα λαμβάνουν πλέον πολύ περισσότερες πληροφορίες με την αυτόματη ανταλλαγή. Ο στόχος λοιπόν αυτής της νομοθεσίας είναι να πιάσουμε τη φορο ε, διαφυγή, να υπάρχουν οι καταλληλοί και οι φορολογικές διοικήσεις σε πολλές χώρες και στη δικιά μου έχουν υποφέρει από περικοπές προσωπικού και θα ε, θεωρούμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το Κετσιαδής δεν κάνει το λόγο, Μπαρμπαρα Κάπελ δεν βλέπω. Κύριε Μορέλ, έχετε τον λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε του συναδέλφους και χαίρομαι πραγματικά που βλέπω ότι ως προς τον πολιτικό στόχο που είναι να τερματιστούν κάποιες πρακτικές και για να χρησιμοποιήσω και τη φράση του συναδέλφου από τους πράσινους να βρεθούμε πραγματικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη γραμμή κατά της φορολογικής επιθετικής βελτιστοποίησης συμφωνούμε όλοι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ως προς τον πολιτικό αυτό στόχο υπάρχει σύγκληση απόψεων. Προφανώς θα γίνουν κάποιες ε, συζητήσεις όσον αφορά την ανδρομική ισχύ Νοέμβριος 93, ε, μα εδώ χρησιμοποίησα την έναρξη της συνθήκης του Μάστριχτ και ουσιαστικά τους νέους κανόνες για την κυκλοφορία των κεφαλαίων σε σχέση με τρίτες χώρες. Καταλαβαίνετε πάντως ποιος είναι ο απότερος στόχος. Αν περιοριστούμε μόνο στα μελλοντικά φορολογικά τεχνάσματα και στις μελλοντικές φορολογικές ρυθμίσεις, χάνουμε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του προβλήματος, ότι έχουμε συσσωρεύσει ένα τεράστιο αριθμό τέτοιων φορολογικών διευθετήσεων, τις οποίες θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά τώρα το εμπορικό απόρριτο, ας μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα μιλάμε για πληροφορίες που πηγαίνουν μόνο και αποκλειστικά προς φορολογικές αρχές. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν τα στοιχεία αυτά αλλού. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υφίσταται για κάποια απειλή, ότι ε, η υπόλοιψη των επιχειρήσεων κινδυνεύει. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι τα μέτρα αυτά δεν τα θέλουμε μόνο εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά τα περιμένουν και πάρα πολλές επιχειρήσεις και κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρούν ότι ζημιώνονται πάρα πολύ γιατί κατά αναλογία υποβάλλουν πολύ μεγαλύτερο φόρο από ό,τι πολύ μεγαλύτερες τους επιχειρήσεις. Και δυστυχώς αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Επομένως, δεν ταποκρινόμαστε μόνο στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και σε πάρα πολλές επιχειρήσεις που, όπως είπα, θεωρούν ότι το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα δεν είναι δίκαιο. Εκ των προτέρων, λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για τη μελλοντική εργασία που θα έχουμε και είμαι σίγουρος θα καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό και φιλόδοξο αποτέλεσμα, γιατί όπως το είπατε όλοι σας και συμφωνώ με σας, αυτό το οποίο θέλουμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτή να κρατήσει, στον τομέα αυτό να κρατήσει πραγματικά μια στάση υποδειγματική. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, α δούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα. 15 Δεκεμβρίου η, το μεσημέρι είναι η ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών. Στις 11 Ιανουαρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε στις 24-25 Ιανουαρίου στην Επιτροπή μας, ενώ στη δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. που είναι η συζήτηση για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου Ουσιαστικά εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δίνουμε τη σύμφωνη γνώμη μας, μια πρόταση μόνο περιέχει έκθεση, για τη διμερή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση. Όπως ξέρετε, υπεγράφει η συμφωνία αυτή στις 22 Σεπτεμβρίου μετά από πολλούς γύρους διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμοδίων αρχών των ΗΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερωνόταν τακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπουν οι συνθήκες. Ευχαριστούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση αυτή και θα ήθελα και να συγχαρώ, βλέπω και την εκπρόσωπο εδώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να συγχαρώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πολύ θετικό αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εμείς στην έκθεση προτείνουμε να στηρίξουμε, να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας στην διμερή ε, αυτή συμφωνία. Πολύ σύντομα θα ήθελα να συνοψίσω τα σημαντικότερα στοιχεία της συμφωνίας αυτής. Θέλουμε να έχουμε ένα νέο σύστημα όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση και την προληπτική εποπτεία. Δεν θα υπάρχει πλέον αυτή η περίοδος των πέντε ετών που προβλεπόταν, ε, όπου έπρεπε να τηρηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης και αντασφάλισης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών οι διατάξει ήταν πολύ πιο ελαστικέ. επομένω θεωρούσαμε ότι ήταν υπερβολικό το ποσό εγγύησης σε 40 δισεκατομμύρια περίπου, 40 δισεκατομμύρια δολάρια που προβλεπόταν για την ευρωπαϊκή πλευρά. Μέσω της συμφωνίας αυτής επίσης θα καταργήσουμε τις απαιτήσει που προβλεπόταν από κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπάρχει συγκεκριμένη εγγραφή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εταιρεία η οποία θέλει να προσχωρήσει σε δραστηριότητες ασφάλισης και ασφάλισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διατάξεις αυτές λοιπόν, οι απαιτήσει αυτές θα εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση της αντασφάλισης, στην περίπτωση που μιλάμε για ποσά άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων και ουσιαστικά αυτό συνάδει με την ε, νομοθεσία, την σχετική νομοθεσία των ΗΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Αφαρικαιότητα 2. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, πάλι στα πλαίσια της νομοθεσίας ε, Insolvency 2, προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν δραστηριότητα σε τρίτη χώρα Πάλι εδώ πέρα προβλέπεται μία εποπτεία με συγκεκριμένους κανόνες κεφαλαιακών απαιτήσεων στις χώρες εκείνες όπου υπάρχει πραγματική δραστηριότητα. Επομένως, δεν θα ισχύει η προϋπόθεση αυτή για τις αμερικανικές εκείνες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς όμως τα κέρδη να πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκή επικράτεια. Τέλος, ένα σημαντικό επίτευγμα έχουμε και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών αρχών, η αυξημένη ροή πληροφοριών μεταξύ των δύο πλευρών θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε επικαλύψεις, να αποφύγουμε να συλλέγουμε τις ίδιες πληροφορίες δύο φορές και θα έχουμε και καλύτερη συμμόρφωση με τους κανόνες περί απορρίτου. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να οδηγηθούμε σε ένα καλύτερο μνημόνιο συνεννόησης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υποπτικών αρχών των Ευρωπαϊκών και των Αμερικανικών. Εν γέννη, όπως υπόθηκε ήδη, θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή είναι ιδιαίτερα θετική. Συγχαίρω για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώς η πρόταση του υποφαινόμενου είναι να δώσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη σύμφωνη γνώμη μας για τη συμφωνία αυτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλάμε για μια διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Επομένως, δεν μπορούμε εμείς να τροποποιήσουμε την, το περιεχόμενο της πρότασης, μπορούμε απλώς να πούμε ναι ή όχι. Εμείς από ό,τι θα ψηφίσουμε στις 24-25 Ιανουαρίου του 2018, την ίδια μέρα δηλαδή που θα εξετάσουμε και τις τροπολογίες. Ο κύριος Μπάλτς τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετίζω την συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ και ευρωπαϊκή Ένωσης και έτσι διασφαλίζουμε ότι τα μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εταιρείες αντασφάλισης ε, που μιλάμε για ύψος 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήπα θα πρέπει να μειωθούν τα επόμενα χρόνια. Έτσι αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αντασφαλιστριών εταιριών σε διεθνές επίπεδο και θεωρώ ότι έτσι ωφελούνται και οι δύο πλευρές. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι θετικό το ότι η Κομισιόν συχνά θα κάνει άτυπες ενημερώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις ε, διεθνείς ε, συμφωνίες όταν μιλάμε για την διεθνή εποπτεία. Όμως εδώ πέρα θεωρώ πως ε, είχε η Κομισιόν καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ξεκάθαρα. Συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύμφωνης γνώμης ε, και να στείλουμε ένα μήνυμα για μια διεθνή παροχή υπηρεσιών, ε, ένα μήνυμα υπέρ της διατλαντικής συνεργασίας. Εγώ γύρισα σήμερα το πρωί από την Ουάσιγκτον, ε, κάνα μια επίσκεψη κάποιων ημερών με την αντιπροσωπεία για είπα και βέβαια στην διατήρηση, διατήρηση ανοιχτών αγορών. Οπότε η ομάδα μας συμφωνεί ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω κάποιον να τον σκιωδησηγηθεί, οπότε μπορούμε να δώσουμε τώρα τον λόγο αν, αν έχετε κάτι να πείτε έτσι. Κάτι σύντομο συγκομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την θετική σας ε, θέση στην πολύ σημαντική αυτή συμφωνία, όπως ε, σωστά είπε ο κύριος Μπάλτς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την θέση των ευρωπαϊκών αντασφαλιστικών εταιριών που έχουν μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής αγοράς ασφαλιών και έτσι θα έχουν ακόμα περισσότερα στη σημαντική αυτήν αγορά. Είμαστε στη διάθεσή σας βεβαίως ανα πάσα στιγμή για να ενημερώσουμε την ΕΚΟΝ και το Κοινοβούλιο για οποιοδήποτε ερώτημα πιθανώ έχουν για την συμφωνία και την εφαρμογή της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα, 14 Δεκεμβρίου οι τροπολογίες ε, και θα ε, δούμε και την ίδια μέρα, στην ίδια συνεδρίαση. Τη συνεδρίαση μας τον Ιανουάριο. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ. Και τα λέμε στο Στρασβούργο, ε, όλος εξαιρετικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεδρίαση.